Buonasera a tutti. Allora, iniziamo con... Ας αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Έχετε την ημερίση, το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, επειδή έχετε μοιραστεί το κείμενο, θεωρούμε ότι εγκρίθηκε. Ο μεγαλύτερος, ο πιο πολύς χρόνος μας σήμερα και αύριο θα είναι για τις ισπανικές αναφορές στο δικαίωμα πνευματικής διευθυνσίας ως προβλέπει ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παρούσα η κυρία Λίτσα Μπανσαντολίνη, Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου για το Περιβάλλον, υπεύθυνη για τις ακτές, που μας το όρισε, μας όρισε ως συνομιλητή μας η Ισπανική κυβέρνηση χαιρετίζει τον κυρία Πας Σαντολίν. Παρίστανται επίσης οι εκπρόσωποι των περιφερειών. Έχω ε, δεν έχω τα ονόματα, τους χαιρετίζω αν είναι παρόντες. Όπως επίσης και πολλούς από τους ετούντες που είναι παρόντες για να παρακολουθήσουν τη συζήτηση, αλλά θα τους δώσω το λόγο αύριο. Σήμερα το απόγευμα στη συνεδρίασή μας συμμετέχουν και τέσσερα μέλη από τη Γερμανική Βουλή, τους οποίους επίσης ο κύριος Γιούντερ, η κυρία Γιώνας, ο κύριος Τίπερ και η κυρία Χάρτσερ. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας συνεδρίαση. Επίσης παρίστανται και οι, οι ετούντες 0058 11.43 κύριοι Σάνιτας και 1120 2009 Μάρκο Γκριφίνη Φυσικά υπάρχει ο κατάλογος των αναφορών που θα πρέπει να ξανανοίξουμε να κλείσουμε με την αιτιολόγηση και αυτό έχει μοιραστεί ήδη από την περασμένη εβδομάδα. Δεν υπήρξαν ενστάσεις ή σχόλια. Άρα, οι συστάσεις στο κείμενο αυτό θεωρούνται και αυτές εγκεκριμένες. Τελευταία ανακοίνωση. Η συνεδρίαση της επιτροπή μας που για 7 και 8 Απριλίου, επειδή οι περισσότεροι συνάδελφοι το ζήτησαν, αναβάλλεται για 26 και 27 Απριλίου. Ας έρθουμε τώρα στις αναφορές. Πρώτη, η ακρόαση των Ισπανικών αρχών σχετικά με τις αναφορές για τον νόμο περί των ακτών. Γι' αυτό και θα δώσω το λόγο αμέσως στην εκπρόσωπο της Ισπανικής κυβέρνησης. Buenas tardes. Eh, presidente. Καλησπέρα σα, κύριε και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη τη Επιτροπή των Αναφορών. Θα ήθελα καταρχήν να σα ευχαριστήσω για την ευκαιρία που δίνετε στην Ισπανική κυβέρνηση να έρθει και να μιλήσει της Επιτροπή σας, στην Επιτροπή σας δίνοντας κάποιες έστω και σύντομες εξηγήσεις για τις αρχές που διέπουν τον νόμο περιακτών και τους στόχους αυτής της νομοθεσίας και να σας εξηγήσουμε τους θεμελιώδεις ορισμούς αυτού του νομοθετήματος αποσαφηνίζοντας κάποιες ιδέες που παρεξηγήθηκαν. Επίσης θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω ποια είναι η πρακτική που χρησιμοποιήθηκε και που δημιούργησε προβλήματα. Κάτι που είναι γνωστό σε όλους, γι' αυτό και δεν θα επιμείνω πολύ σε αυτό. Καταρχήν θα ήθελα να σας ε, πω για ποιους λόγους σχεδιάσαμε αυτό το νόμο περί ακτών, περί γιατί είναι απαραίτητος για να προστατεύσουμε τις ε, Ισπανικές ακτές. Οι Ισπανικές ακτές ε, έχουν γνωστές περιβαλλοντικές αξίες ε, και Ιδηλιακό τοπίο. Επίσης, ε, πολυμορφία από άποψη χλωρίδας και πανίδας. Πολύ σημαντική βιοπικιλότητα που θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Μετά από διάφορα γεγονότα, γνωρίζουμε ότι οι κλιματικές αλλαγές απειλούν τις ακτές. Το ίδιο και οι θεομηνίες και διάφορες φυσικές καταστροφές. Επίσης, συνιστούν σημαντικές απειλές για τις ακτές οι ακτές έχουν οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική αξία, αλλά και αξία αναψυχής. Σημαντική ψυχαγωγική αξία που υφίσταται ταυτόχρονα τεράστιες πιέσεις, γιατί θα πρέπει να συμφιλιώσουν περιβαλλοντικές αρχές με άλλες πιέσεις που πολλές φορές προκύπτουν από την ανθρώπινη δράση, από ανθρωπογενείς παράγοντες και θα πρέπει να γίνει αυτή η συμφιλίωση, να βρεθεί αυτή η ισορροπία. Η νομοθεσία αυτή είναι από το 1988 σε ισχύ, ισχύει δηλαδή πάνω από 20 χρόνια και έχει τρεις βασικές πτυχές ως προς το περιεχόμενό της. Καταρχήν, η νομοθεσία αυτή περιλαμβάνει τη ρύθμιση του δημόσιου θαλάσσιου και χερσαίου χώρου. Πρόκειται για ένα στοιχειώδες και κλασικό νόημα της νομοθεσίας μας που προβλέπει ότι ένα τμήμα των αγαθών ανήκουν στην κρατική περιουσία. Δεύτερον, η νομοθεσία αυτή προβλέπει κάποιους περιορισμούς ακριβώς εξαιτίας τη ανάγκης προάσπισης αυτού του ευαίσθητου χώρου που είναι οι ακτέ, προβλέπει λοιπόν μια σειρά περιορισμών στη δυνατότητα ε, εξάπλωσης της ε, πολεοδομίας σε μια πολύ στενή ζώνη που σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή θέλει να αποφύγει κάποιες ε, πολεοδομικές υπερβολές. Επίσης προβλέπει κάποιες ε, εξουσίες των τοπικών και περιφερειακών αρχών που προβλέπουν ε, κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις ώστε τα σχέδια τα πολεοδομικά και τα ρημοτομικά να γίνονται σεβαστά. Στη συνέχεια θα σας εξηγήσω τι στη δημόσιος χώρος και ποιες είναι οι ρυθμίσεις και οι περιορισμοί της ιδιωτικής περιουσίας εξαιτίας του δημόσιου χώρου. Καταρχήν, για να δούμε ποιο είναι το πεδίο εφαρμογή ε, του νόμου περί Λου του 1988. Όπως βλέπετε αριστερά, έχουμε την έννοια της ε, κρατικής ε, περιουσίας ή του δημόσιου χώρου και αριστερά έχουμε τις δουλειές ή τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε, αυτό το δημόσιο, σε αυτή τη δημόσια περιουσία, στην κρατική περιουσία. Τι είναι κρατική περιουσία. Όπως σας είπα, ο όρος της κρατικής περιουσίας έχει παράδοση στην Ισπανία. Μακρόχρονη παράδοση. Μακραίωνη θα έλεγα. Και είχαμε ανέκαθεν έναν γυαλό μία ακτογραμμή που θεωρούνταν ε, κρατική περιουσία. Το Σύνταγμά μας, ακολουθώντας αυτή την παράδοση, το 1978, το Ισπανικό Σύνταγμα το 1978 για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνει ένα νόμο που έχει συνταγματική αξία και που θεωρεί την ακτογραμμή ως κρατική περιουσία, ως κρατικό αγαθό. Και μάλιστα αυτή η κρατική περιουσία εξορισμού θα πρέπει να χρησιμοποιείται ελεύθερα, δημόσια και δωρεάν από όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η βασική αρχή που διέπει τη χρήση αυτών των ακτών. Και η έννοια της κρατικής περιουσίας και της ε, δυνατότητας συλλογική χρήσης από τους πολίτες ε, ουσιαστικά αντιβαίνει στην αρχή ιδιωτικής περιουσίας στις ακτογραμμές, στις ακτές. Και για να ξέρουμε γιατί μιλούμε, γιατί περιουσιακά στοιχεία μιλούμε και γιατί ε, θέλουμε τέτοια προστασία. Ουσιαστικά μιλούμε για τις ακτές, για τις Αθήνες, για τις υγρές ζώνες, για τους βάλτους, για τις ζώνες που βρέχονται από τα κύματα. Αυτά είναι όλα τα τμήματα που εμπίπτουν στον στο νόμο περί του 1988 που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Όλα αυτά τα, όλες αυτές οι γεές είναι ε, ιδιωτικές, όταν είναι ιδιωτικέ δεν αλλάζει το καθεστώς της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά προβλέπονται κάποιοι περιορισμοί σε αυτή την ιδιωτική περιουσία και κυρίως ε, απαγόρευση οικοδόμησης κατοικιών. Αυτή είναι η ουσιαστική απαγόρευση, ο βασικός περιορισμός σε, αυτές τις, ε, σε αυτά τα ιδιωτικά ακίνητα και μάλιστα συνήθως ε, η δουλεία προστασίας αφορά τα 100 μέτρα, δηλαδή ε, περιοχές, ε, ακίνητα που βρίσκονται δίπλα στην ε, κρατική περιουσία και είναι ιδιωτικά, δεν μπορούν ε, πέρα από τα 100 μέτρα, πιο κοντά από 100 μέτρα από τη θάλασσα να κατασκευάζουν οικίες. Και μάλιστα μετά την νομοθεσία του 88 από τα 100 μέτρα περάσαμε στα 20. Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε τον αντίκτυπο της κατασκευής σε μια πολύ ευαίσθητη ζώνη που είναι οι ακτές, οι αμοθήνες, ε, κάποιοι υγροβιότοποι κοντά στις θάλασσες και ούτω καθεξής. Τώρα πώς γίνεται αυτή η οριοθέτηση. Και ερχόμαστε αυτό στο, σε αυτόν τον όρο της οριοθέτησης, που είναι μια διοικητική διαδικασία που διαχωρίζει την κρατική περιουσία από την ιδιωτική περιουσία. Και μάλιστα καθορίζει το εύρος αυτής της λωρίδας της ε, προστασίας. Η έγκριση αυτής της οριοθέτησης και ο νόμος περί Αγιαλού υπεριακτών εφαρμόστηκαν από τη θέση ισχύ του νόμου περιακτών το 1988. Και εδώ βλέπετε ε, την εξέλιξη των διαφόρων χιλιόμετρων οριοθέτησης που υιοθετούνται κάθε χρόνο από το 1988 μέχρι σήμερα. Όπως βλέπετε πρόκειται για σταδιακή εφαρμογή αυτής της οριοθέτησης και από το 2004-2005 ελάχιστη είναι η πρόοδος που σημειώθηκε. Αυτή η διαδικασία της οριοθέτησης, δεσιλίνδε προβαίνει στο διαχωρισμό στην οριοθέτηση μεταξύ της κρατικής και της ιδιωτικής περιουσίας. Και νομίζω ότι αυτή η διαδικασία που έχει κατά μέσο όρο ισχύει διετή είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και πολύ επίπονη γιατί προβλέπει τεχνικές μελέτες, ε, μελέτες εμπειρογνωμόνων, μια διαδικασία προσφυγής από τους ε, ενδιαφερόμενους. Επίσης, αν κάποιος ιδιοκτήτης ε, εκφράσει σχετική αίτηση, γίνεται μια επιτόπου πραγματογνωμοσύνη από τους εκπροσώπους της πολεοδομίας για να γίνει μια επιτόπου εξέταση αυτής της οριοθέτησης. Και μάλιστα προβλέπεται και δυνατότητα προσφυγής κατά της ε, οριοθέτησης ε, στα διοικητικά δικαστήρια. Τουλάχιστον αναγνωρίζεται σε δύο βαθμούς η προσφυγή. Υπάρχει λοιπόν έλεγχος και διοικητικός αλλά και δικαστικός και μέσω των πολιτικών δικαστηρίων και κατοχυρώνεται το δικαίωμα προσφυγής κατά των πράξεων οριοθέτησης. Να δούμε τώρα πώς προβλέπεται η εφαρμογή αυτής της οριοθέτησης και ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της οριοθέτησης για τι οικίε, ή τα κτίσματα είτε της κρατική είτε της ιδιωτική περιουσία. Ό,τι αφορά την κρατική περιουσία, βλέπουμε καταρχήν αν τα κτίρια αυτά ήταν νόμιμα ή αυθαίρετα. Αν μια κατασκευή είναι νόμιμη, έχει την πολεοδομική άδεια, τις απαραίτητες προσημειώσεις και μεταγραφές, μετατρέπουν το δικαίωμα κυριότητας σε δικαίωμα χρήσης και επικαρπίας που μπορεί να φτάσει μέχρι και 60 χρόνια. Και μάλιστα το δικαστήριο που έκρινε κατά πόσο είναι συνταγματική αυτή η διάταξη δήλωσε ότι αν γίνεται απαλωτρίωση ενός ιδιωτικού δικαιώματος, δικαιώματος ε, ακινήτου, θα πρέπει να εξεταστεί το ύψος της αποζημίωσης. Αν η αποζημίωση αυτή που δίνεται για τα 60 χρόνια είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Αυτό εξετάζει το δικαστήριο. Σε περίπτωση που ήταν δίκαιη αποζημίωση, το δικαστήριο έκρινε ότι από τη στιγμή που η παλωτρίωση συνοδεύεται από δίκαιη αποζημίωση και ισορροπημένη, γίνεται σεβαστό το δικαίωμα της κυριότητας. Αυτά για τις ε, νόμιμες κατασκευές. Τώρα για τα αυθαίρετα και μάλιστα αυθαίρετο θεωρείται ένα κτίσμα, παράνομο δηλαδή, αν χτίστηκε χωρίς πολεοδομική άδεια, αυτή που απαιτούνταν, ή αν δεν συνοδεύεται από τους απαραίτητους τίτλους ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση αυτή, αν πρόκειται για τέτοιες κατασκευές, χωρίς πολεοδομική άδεια, αυθαίρετες ή χωρίς νόμους τίτλους, ξεκινάει μια διαδικασία μια χαρακτηρισμού αυτού του αυθαίρετου ως ε, κτίσματος που αντιβαίνει στον νόμο περιακτών και μάλιστα με δυσμενείς περιβαλλοντικές συνέπειες. Εδώ έχουμε ορισμένα παραδείγματα τέτοιων δράσεων, αυθαίρετων κτισμάτων, για να δείτε πώς ήταν η προηγούμενη κατάσταση και πώς ε, η κατάσταση μετά τη δράση που ανέλαβε η Ισπανική κυβέρνηση για την εξάλληψη αυτών των κτισμάτων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κτίσματα που έγιναν στο, στη ζώνη δουλείας ε, της ε, ιδιωτικής περιουσίας, προσπαθήσαμε να αφήσουμε την κατάσταση όπως υπήρχε και πριν το νόμο του 88, δηλαδή εξακολουθούν να θεωρούνται ιδιωτική περιουσία αυτές οι ζώνες, μπορούν οι ιδιοκτήτες τους ε, να κάνουν κάποιες βελτιώσεις ε, στις ζώνες αυτές, αλλά δεν μπορούν να ανεγείρουν νέα κτίσματα. Και πρόκειται για ιδιωτικές περιουσίες που σας ε, επαναλαμβάνω που είναι όμορες κρατικής περιουσίας στις ακτές. Αυτές ήταν ε, οι βασικές αρχές που διέπουν τον νόμο περιακτών και βασικός μας στόχος ήταν η προάσπιση του περιβαλλοντικού παράκτιου τμήματος και της αποφυγής ε, αντιπεριβαλλοντικής δράσης και των κατασκευών στις παράκτιες ζώνες. Αυτές ήταν ε, οι βασικές αξίες και οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται με τον νόμο περιακτών. Ευχαριστώ. Grazie Σας ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγή. Θα δώσω αμέσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν και μετά στους συναδέλφους. Πρέπει να δώσει απάντηση η Κομισιόν. είτε θα επιβεβαιώσει τις καταγγελίες των αναφορών, διότι οι αναφερόμενοι με πάρα πολλές αναφορές αναφέρονται συγκεκριμένα σε παραβάσεις των συνθήκων οδηγιών της Ένωσης βασικών αρχών που εμπεριέχονται στις συνθήκες ή που υπάρχουν στην θεμελιώδη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, και στην Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΕΣΔΑ. Και επισημαίνω τα εξή δύο τεινά στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. σχετικά με την αρμοδιότητα εμεί των κοινωτικών οργάνων να παρέμβουν. Είναι ο μεγάλος αριθμός περιπτώσεων που έχουν αναφερθεί σε μας. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ατομικές παραβάσεις, επιμέρους εξαιρέσεις παραβάσεις, άρα δεν, αφαιρούν, δεν αφορούν τα κοινωτικά όργανα πρέπει να τα δούμε ως κάτι το γενικό, γενικές περιπτώσεις, Δηλαδή, επαναλαμβάνω αφορούν πολυπληθείς αναφερόμενους και όχι μόνο Ισπανούς ε, υπηκόους αλλά και Ευρωπαίους υπηκόους γενικότερα. Έχουμε Ολλανδούς, Γάλλους, Γερμανούς και από άλλες χώρες της Ένωσης. Και το δεύτερο σχετικά με το πόσο είναι αρμόδιοι ή όχι τα κοινοτικά όργανα να παρέμβουν, δεν μπορούν να παρέμβουν αν κατά κάποιο τρόπο δεν τίθεται να αμφιβόλει το κοινοτικό δίκαιο. Από τη στιγμή που στις συγκεκριμένε περιπτώσεις υπάρχει πρωτεύουσα χρήση κοινοτικών κονδυλίων που δαπανώνται στις χώρες μέλη με βάση εφαρμογή μια συγκεκριμένη κοινοτική νομοθεσία μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι μιλάμε για θέματα που όντως ε, αφορούν το κοινοτικό δίκαιο. Και τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχεδόν απαντήσατε. Μ' ακούτε καλύτερα τώρα. Σχεδόν απαντήσατε στην ερώτηση που με έγινε μόνος, ε, μόνοι σας, διότι ξέρετε από προηγούμενες αναφορές ότι το βασικό πρόβλημα είναι πρόβλημα νόμου περί ακινήτων. Επανειλημμένα έχουμε πει στην Επιτροπή σας, δυστυχώς, ότι αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, όταν υπέβαλε πέρσι το Φεβρουάριο την γνωμοδότησή της στην Επιτροπή σας για το θέμα αυτό, σας παρέπεμψε στην ε, νομολογία στην υπόθεση Ανιπέλη, όπου το δικαστήριο είπε πολύ καθαρά ότι το θέμα του νόμου περί και των απαλωτριώσεων δεν είναι καθόλου αρμοδιότητα κοινοτική, που δεν ήθελαν καν να υποβάλουν γνωμοδότηση προς τον Ιταλό δικαστή που παρέπεψε την υπόθεση στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όσον αφορά τη Γενική Αρχή, κυρία Πρόεδρε, ξέρω ότι αυτό είναι απογοητευτικό. Δεν έχουμε δυνατότητα, δεν έχουμε τη νομική βάση για να παρέμβουμε. Όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση λοιπόν, το αν αυτές οι μεμονωμένες υποθέσεις που ε, ουσιαστικά καταλήγουν ε, ε πρακτική κατ' δεν ε, είναι ένα θέμα που να μπορούμε να ε, συζητήσουμε. Όσον αφορά τους κοινοτικούς πόρους, τη δεύτερη σας ερώτηση, όσον αφορά τις απαλωτριώσεις που ανέφερα, Εγώ δεν έχω δει σε καμία από τις αναφορές που υπέβαλαν, που, που υπευλήθησαν ε, χρήση κοινοτικών πόρων. Τα διαστροτικά ταμεία η Κομισιόν ήταν πάντα κατά τη χρήση διαρθρωτικών ε, ε, ταμείων και κοινοτικών πόρων για απαλωτριώσει. Γι' αυτό, για παράδειγμα, στις, συμβάσει συμβάσεις για ε, οδικές κατασκευές, πολύ μικρό ε, κομμάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποζημιώσει σε, σε περίπτωση απαλωτρίωση. Σε μία από τις αναφορές που έχετε στην ημερήσια διάταξη, Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι ε, κοινοτικό πρόγραμμα οδήγησε σε διάβρωση των ακτών λίγο πιο κάτω, το οποίο σημαίνει ότι ε, ακίνητα που παλιά ήταν σε ασφαλή απόσταση από τις ακτές, ε, λόγω της διάβρωσης των ακτών έφτασαν πολύ κοντά στην ακτή. Και αυτό είναι πολύ δυσάρεστη κατάσταση για τον αναφέροντα είναι όμως με μονομένη περίπτωση που δεν νομίζω ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να γενικεύσουμε για να βγάλουμε πιο γενικά συμπεράσματα όσον αφορά την ε, χρήση των πόρων μας. Όσον αφορά τη δραστηριότητα στις παράκτιες περιοχές, ε, πρόσφατα υποβάλαμε στο Συμβούλιο, φέτος δηλαδή το Γενάρη, πρόταση η κοινότητα να υπογράψει πρωτόκολλο για την διαχείριση των ακτών της ε, Σύμβασης της Βαρκελόνης. Αυτή η σύμβαση είναι μια διεθνή σύμβαση του 1970 για την προστασία της Μεσογείου. Πρόσφατα ε, προστάθηκε ένα πρωτόκολλο στη σύμβαση αυτή για την προστασία των ακτών που περιέχει χρήσιμες διατάξεις ε, διαφάνειας ε, και ε, σωστής διαδικασίας για το κοινό όσον αφορά τη διαχείριση παράκτιων περιοχών. Η Ισπανία δεν έχει επικυρώσει ακόμα το πρωτόκολλο αυτό, αναμένεται όμως να το κάνει εντός της φετινής χρονιάς. Προς ενημέρωσή σας έχουμε φέρει αντίγραφα της πρότασης της Κομισιόν προς το Συμβούλιο να συνυπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση την, το πρωτοκόλλο αυτό κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Ε, το έχουμε στα Ισπανικά, Ιταλικά, Αγγλικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Και αρχίζει η συζήτηση. Καλό τους συναδέλφους να μην μακρηγορούμε γιατί ήδη δέκα έχουν ζητήσει το λόγο. 11. Έλμερ πρώτος. Κύριε Πρόεδρε. Θυμάμαι όταν χώρε θέλουν να μπουν στην Ένωση, ένα όρο, είναι να έχουμε οικονομία τη αγορά που να λειτουργεί σωστά. Και προπόθεση μια τέτοια οικονομία τη αγορά είναι κράτο δικαίου, δικαιώματα ιδιοκτησία και τα συμβόλαια να είναι νόμιμα και να εφαρμόζονται. Εδώ αυτό δεν ισχύει στην Ισπανία. Και πιστεύω η Ισπανία αν ήταν εκτό Ένωση σήμερα και έκανε αίτηση για ένταξη θα είχε σοβαρό πρόβλημα. Ακούσαμε πάρα πολλά από το Υπουργείο για το πόσο περίπλοκο είναι αυτός ο νόμος περί ακτών ή αλλού, αλλά ουσιαστικά τα δικαιώματα ιδιοκτησία και τα συμβόλαια των πολιτών στην πραγματικότητα βάζουν στην πάντα. Ένα παράδειγμα που σήμερα το έμαθα στην Καταλωνία, σε μια περιοχή, η περιοχή των ακτών επαναορίστηκε από την ακτή για να συμπεριληφθεί μια μαρίνα που ήταν εκεί χρόνια. Τώρα και όλα τα ε, ό,τι είχε σχέση με τη μέρα αυτή επαναδιορίστηκαν ως της ακτής και όλη αυτή η μονάδα με εκατοντάδες περιουσίες, πολλά ιδιοκτησία υπηκών της Ένωσης, ξαφνικά υπάρχει κίνδυνος να υποστούν ε, απαλωτρίωση. Εγώ, κατ' επανάληψη στο παρελθόν, έχω πάρει δεκάδες επιστολών, πολύ συγκινικών, πολλά από την πατρίδα μου, αλλά το ίδιο νομίζω ισχύει και για άλλους συναδέλφους. Ε, κάποιος βγαίνει στη σύνταξη, ε, επενδύει στην Ισπανία Φερρυπίν, κάνει όλα τα σωστά που πρέπει να κάνει, παίρνει ντόπιου δικηγόρους και μετά από μήνες ή χρόνια ξυπνάνε μια μέρα και ξαφνικά βλέπουν μπουλτόζες στην πόρτα τους και ένα ένταλμα απαλωτρίωσης ή έξωσης. Αν είχε γίνει κάτι τέτοιο στη χώρα μου, Πιστεύω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί θα θέλουν να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα και θα το έκαναν για να προστατεύσουν τα δικαιώματα των πολιτών. Και απογοητεύομαι πάρα πολύ για το ότι πολλοί Ισπανοί συνάδελφοι, από ό,τι βλέπω, θέλουν να προστατεύσουν κυρίω την Ισπανική κυβέρνηση, του ντόπιου πολιτικού, τοπική αυτοδιοίκηση, δήμαρχου, εργολάβου. Ακούμε ένα σωρό ιστορίε για διαφθορά μεταξύ όλων αυτών των ατόμων. Αποτέλεσμα, όλη αυτή η σειρά των ε, γεγονότων αυτών βλάπτει και το κύριο της Ισπανίας αλλά και την αγορά κινήτων στην Ισπανία. Με ρωτήσει κάποιος να αγοράσει στην Ισπανία. Η πρώτη μου αντίδραση είναι όχι, μην αγοράζει στην Ισπανία. Κάνω έκκληση λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, στην Κομισιόν. Άκουσα τη θέση της Κομισιόν για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, αλλά τα δικαιώματα στην ιδιοκτησία και η εφαρμογή των συμβολέων είναι βασικός στυλοβάτης της ελεύθερης αγοράς με βάση την οποία λειτουργεί η Ένωση. Και είναι απαράδεκτο η Ισπανία να παρακάμπτει αυτούς τους νόμους, παραβιάζοντας νόμους πολιτών και της χώρας μου και από πολλές άλλες χώρες και από την ίδια την Ισπανία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σα παρακαλώ όχι τέτοιου είδου συμμετοχέ, γιατί θα έχουν δυσκολίε στο να συνεχίσουμε έτσι. Μάτω Αντρογκάρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από λίγο, μετά την ομιλία του εκπροσώπου, της εκπροσώπου της κυβέρνησης Ισπανίας, είπε κάποιος από τους αναφέροντες ότι μας έδωσαν ε, μία διάλεξη για οριοθέτηση και δημόσιο κτήμα ε, για να μας απαλωτριώσουν ε, οικίες που είναι οικογενειακή περιουσία εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Νομίζω ότι οι καταχρήσει αυτού του νόμου υπερβαίνουν το θέμα του δικαιώματος ιδιοκτησίας και την ε, εφαρμογή μιας νομοθεσίας. Μιλούμε για ανθρώπους που έχουν περάσει χρόνια ολόκληρα σε μια κατοικία, στο Τσοβίτο για παράδειγμα, που χάνουν τα σπίτια τους. Στην περίπτωση του παραρτήματος 2, στο Σαν Παρτολομέ, άνθρωποι χάνουν τα δικαιώματά τους, ενώ είχαν δικαιώματα κυριότητας και μάλιστα δημεύονται ή απολωτηρώνουν την περιουσία τους χωρίς καμία δικαιολογία. Πώς εφαρμόζεται με αναδρομική ισχύ ε, αυτός ο κανόνας, γιατί όταν χάνουν ε, άνθρωποι δικαιώματα που είχαν 300 χρόνια, υπάρχει αναδρομική ισχύ, μην μου λέτε όχι. Επίσης, πώς μετατρέπεται το δικαίωμα κυριότητας σε δικαίωμα ε, προσωρινής ε, χρήσης, που μπορεί μερικές φορές και μέσα σε ένα χρόνο να ανακληθεί. Το ανώτατο δικαστήριο μίλησε για ισορροπημένη και δίκαιη εφαρμογή. Δεν είναι ισορροπημένη και δίκαιη εφαρμογή να ε, αμυφθεί κανεί ή να αποζημιωθεί για ένα χρόνο. Θα πρέπει να αποζημιώνεται για, για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. Και μάλιστα η ίδια κυβέρνηση θα πρέπει να πει. Θεωρεί ότι έχουν αποζημιωθεί δίκαια όλοι αυτοί οι θυγόμενοι από την εφαρμογή του νόμου περί ακτών. θεωρεί η Ισπανική κυβέρνηση ότι προσπίστηκαν τα δικαιώματα κυριότητας και ιδιοκτησία τους. Τι θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θέλουν μια νομική ασφάλεια και όχι μια αυθαίρετη εφαρμογή του νόμου. Αυτό ζητούμε και αυτό θα, θα απαιτήσουμε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάσμαν. Κύριος Κάσμαν. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ε, Ω που συμμετείχα, που, που ηγήθηκα αποστολή στην Ισπανία για το θέμα αυτό, ε, πρέπει να πω ότι ε, περιέργως συμφωνώ διότι είναι... Ε, ε, συντηρητικός πολιτικός, ε, αλλά συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα είπε ο κύριος Χέλμερ. Ε, η κατάσταση αυτή συνεχίζεται από το 2004 χωρίς καμία επίλυση του προβλήματος για τους αναφέροντες, για τους πολίτες της Ισπανίας που ήδη αγόρασαν νόμιμα ακίνητα και ανακάλυψαν ότι δεν υπήρχαν άδειες για τα ακίνητα αυτά. Για αυτούς που, ε, από τους οποίους ε, απαλωτριώθηκαν τα ακίνητα δεν υπήρχε καμία σωστή αποζημίωση και φοβάμαι ότι αυτό έχει ε, μειώσει την εμπιστοσύνη όχι μόνο στην, στον τομέα της ε, οικοδόμησης στην Ισπανία αλλά και στην Ισπανία γενικά. Γι' αυτό παρά τα όσα λέει η Κομισιόν, ε, συμφωνώ με τον κύριο Χέλμερ, συμφωνώ με τον προλαλήσαντα, το θέμα είναι η εφαρμοσιμότητα των των ε, συμβάσεων, ε, τα θέματα της δέουσας επιμελητίας ε, και το θέμα της σωστής νομιμής αποζημίωσης. Κανένα από αυτά τα θέματα δεν έχει λυθεί, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια ευκαιρία. Εάν λέμε ότι μπορούμε να έχουμε ένα νόμο για τις ακτές, θα πρέπει να έχουμε ένα νόμο για το σύνολο της Ισπανίας,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 ε, κατά την εκπόνηση της εκθεσής μου είπε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το νόμο. Ε, δηλαδή δεν είναι κάτι που έχει ψηφίσει μόνο η Επιτροπή μας. Το σύνολο του Κοινοβουλίου έχει πει ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το νόμο. Ε, η Κομισιόν πάντα προσπαθεί να ξεφύγει. λέει ότι όσον αφορά το αν τα ανθρώπινα δικαιώματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητά Ε, αναφέρεται όμω σαφώ στη συνθήκη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μέρο τη κοινή μα βάση και γι' αυτό το λόγο ε, έχουμε δικαίωμα να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, έχουμε υποχρέωση να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω στην ε, κυρία Πρόεδρε ε, ότι οι αναφέροντες μπορούν να έρθουν όχι μόνο όταν παραβιάζονται οι, οι νόμοι ή τα δικαιώματά τους. ο κόσμος μπορεί να υποβάλει αναφορά σε εμά για οποιοδήποτε θέμα. είναι πολύ ευρύ το φάσμα των αναφορών που μπορεί να υποβληθεί. Έχουμε λοιπόν εδώ σημαντική νομοθεσία η οποία παραβιάζεται από την ε, Ισπανία και μιλώ για τη σύμβαση του ε, που λέει ότι έχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες ε, όσον αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία. Για παράδειγμα, έχουμε ε, αίτηση Χωσέ Ορτέγα 174 του 2008, όπου λέμε ότι δεν του δόθηκαν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα όρια, με τα με τα από οικόπεδα κτλ. Και αυτό είναι σαφής παραδίαση της σύμβασης του άρχους ε, και δεν είναι δικαιολογία το ότι εδώ μιλάμε για ε, ιδιωτικά συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, προσυπογράψει την σύμβαση του Άρχους και ειλικρινά με συγχύζει το ότι η Κομισιόν συνεχίζει να ξεχνάει την νομοθεσία ώρες ώρες ε, πραγματικά συγχύζομαι με την Κομισιόν. Να επανέλθω τώρα στην Ισπανική κυβέρνηση. Είναι εξαιρετικό ο νόμος περί ακτών, αλλά η εφαρμογή του γίνεται αυθαίρετα τελείως. Καταρχήν, από το 1988 μέχρι το 2008 δεν εφαρμοζόταν ο νόμος αυτός, τίποτα δεν γινόταν. Και ξαφνικά με πολύ θόρυβο αρχίζει να εφαρμόζεται ο νόμος αυτό. Ε, ο κόσμο όμω δεν βλέπει πώ μπορεί να λειτουργήσει ο νόμο αυτό. Και ε, αν δούμε την εφαρμογή του νόμου αυτού, βλέπουμε ότι ε, μικρέ καλύβε κρεμίζονται και υπάρχουν ξενοδοχεία όπου ο κόσμο έχει τα πόδια μέσα στο νερό λίγο πολύ. και μπορεί να αναρωτηθεί κανεί γιατί είναι νόμιμα τα ξενοδοχεία αυτά. Μιλάμε για το πόσο ευάλωτε είναι οι Ισπανικέ ακτέ, τον πλούτο τη φύση, την πολιτιστική του σημασία. Συμφωνώ απόλυτα. Όταν όμως εξετάσουμε την πραγματικότητα, η αυτή αυτή είναι μία μόνιμη παραβίαση του εξαιρετικού αυτού νόμου και η αυθαιρεσία αυτή στην εφαρμογή του νόμου είναι θέμα στο οποίο θέλω να μου απαντήσουν οι Ισπανικές αρχές. Είσαστε βέβαιοι, μπορεί να εξετάσει κανείς ποιος έχει πάρει άδεια, ποιος, ποιανού έχει γκρεμιστεί το ακίνητο. Διότι για μας Φαίνεται σαν να υπάρχει πολύ σημαντική ε, ε, διαφορά στη μεταχείριση μικρών και μεγάλων. Και θα ήθελα απάντηση από τις ισπανικές ε, αρχές, όπως είπα, γιατί δεν τηρούν την, τις διατάξεις της σύμβασης του Άρχους σχετικά με την πρόσβαση και τι θα κάνει ε, όσο γίνεται πιο γρήγορα για να ε, πληρώσει τι υποχρεώσει του. Είναι αδύνατον οι πολίτε να παραπονεθούν, να προσφύγουν, εάν δεν έχουν ε, πληροφορίε σχετικά με τη βάση πάνω στην οποία έχει ληφθεί μια απόφαση. Δεν έχει νόημα να μπορεί να πει κανεί ότι μπορεί να πάει κανεί στο δικαστήριο. Δεν μπορεί να πάει κανεί στο δικαστήριο αν δεν ξέρει περί πρόκειται. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε πολλού καλού λόγου να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και θα πρέπει να βοηθήσουμε τους συμπολίτε μας, είτε είναι Ισπανοί, είτε είναι πολίτε άλλων χωρών. Θα πρέπει να έχουν τα ίδια κοινά δικαιώματα, ε, θα πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση όσον αφορά την εξέταση της υπόθεσής του. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω φυσικά τους εκπροσώπους της Ισπανικής Κυβέρνησης στη συνεδρίασή μας και θα ήθελα να κάνω μια σύντομη εισαγωγή πριν υποβάλω μια σειρά ερωτημάτων σε εκπροσώπους της Ισπανικής Κυβέρνησης, μια και έχουμε τέτοια ευκαιρία. Θα πρέπει καταρχήν να αντιληφθούμε ότι η υπόθεση αυτή δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως σύνολο. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι το νόμο περιακτών με όλα αυτά τα θέματα. Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα τη φρούτη, να τα έχουμε όλα εδώ, όλα μαζί. Γιατί άλλο ένα ξενοδοχείο, όπως είπε η κυρία Άουκεν, που χτίστηκε πριν από λίγα χρόνια, δίπλα ακριβώ στη θάλασσα, ή ένας α, μήλος που στη χώρα των Βάσκων κατασκευάστηκε το 16ο αιώνα και είναι πολιτιστικό αγαθό, είναι μνημείο. Δεν είναι το ίδιο ένα αυθαίρετο και ή οικισμοί ψαράδων για παράδειγμα. Δεν είναι το ίδιο ένα αυθαίρετο ή παράνομο κτίσμα με υγρο, υγρότοπους ή αλικές που εδώ και αιώνες ε, υπάρχουν στην Ισπανία. Δεν θα πρέπει λοιπόν να τα βάζουμε όλα στο δυο στο τσουβάλι και είμαστε υπέρ της αποκατάστασης, είμαστε υπέρ της πάταξης παρανομίας και των αυθαιρέτων, αλλά δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε αναδρομικά ένα τέτοιο νόμο και να χαρακτηρίζουμε ε, παράνομα κάτι που ήταν νόμιμο με βάση την προηγούμενη νομοθεσία. Μερικές φορές φαίνεται μεροληπτικός, ιδιότροπος αυτός ο νόμος. Εφαρμόζει διακριτική μεταχείριση και μάλιστα τροποποιεί πολλές φορές τις ε, οριοθετήσεις και μάλιστα ο νόμος αυτός ουσιαστικά έπληξε 400.000 Ισπανούς και αλλοδαπούς αλλά και πολλές επιχειρήσεις γιατί χωρίς ενιαίο κριτήριο επαναπροσδιορίζει τα όρια και εφαρμόζει αυθαίρετα την οριοθέτηση, χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων παράνομα κτίσματα που με τον προηγούμενη νομοθεσία ήταν νόμιμα πολίτες υφίστανται δίμευση των περιουσιών τους, απαλωτρίωση χωρίς δίκαιη αποζημίωση. Γιατί αυτό που κρίνουν ε, είναι μόνο το θέμα του κτίσματος, γιατί ε, υπολογίζουν μόνο το κτίσμα και όχι το ακίνητο που από ιδιωτικό κτήμα γίνεται δημόσιο. Ο νόμος περιακτών ε, ουσιαστικά κρίνει τους ιδιοκτήτες ως καταληψίες. Έτσι τους μεταχειρίζεται, σαν να είναι απλοί καταληψίες και σαν να μην έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και κυριότητας. Σε ό,τι αφορά την αναδρομική ισχύ του νόμου, θα ήθελα να ρωτήσω πώς είναι δυνατόν ένας νόμος του 1988 να καλύπτει νομικές καταστάσεις και νομίμως κτηθέντα δικαιώματα που προηγούνται της ε, έγκρισης του νόμου του 88. Γιατί στερείται από πολίτες τα νόμιμα δικαιώματά τους, χαρακτηρίζοντας δημόσιο κτήμα ιδιωτικές περιουσίες που είχαν νόμιμα κτηθεί ε, με βάση προηγούμενη νομοθεσία του 1880. Θα τηρήσετε το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και το, τη συνθήκη που προβλέπει απαγόρευση για την αειδρομική ισχύ των νόμων σε ό,τι αφορά την αυθαίρετη οριοθέτηση. Γιατί κάνετε οριοθέτηση με zigzag και γιατί επίτηδες χρησιμοποιείτε την zigzag οριοθέτηση για να σώσετε συγκεκριμένα κτίσματα. Γιατί τα κριτήρια που χρησιμοποιείτε για την οριοθέτηση δεν είναι ενιαία, αλλά διαφορετικά. Και μια και βρεθήκατε στη συνεδρίαση, θα πρέπει να δώσετε και μια νότα ελπίδας προς τους ετούντες. Σήμερα ακούμε εσά και αύριο θα ακούσουμε του ε, ετούντε στην Επιτροπή Αναφορών. Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση για να επιλύσει τα προβλήματα που ακούσατε σήμερα στην Επιτροπή. Τι πρόκειται να κάνει η Ισπανική κυβέρνηση για να θέσει ένα τέρμα σε αυτή την ανασφάλεια δικαίου που έχει δημιουργηθεί, σε αυτή την έλλειψη τη βεβαιότητα δικαίου εξαιτία των δράσεών σα Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τουργκάη, ο κύριο Μέγερ. Σα ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα κυρία Πρόεδρε να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Ισπανικής Κυβέρνησης για την παρουσία της στη συνεδρίασή μας και να ευχαριστήσω θερμά και τους ετούντες που μας δίνουν την ευκαιρία να εξετάσουμε ένα θέμα που ενδιαφέρει ένα πολύ σημαντικό τμήμα των ε, Ευρωπαίων πολιτών, είτε είναι Ισπανοί είτε είναι ε, πολίτες άλλου κράτους. Εγώ είμαι υπέρ του νόμου περί ακτών και αλλού, αλλά δυστυχώ ε, διαπιστώνουμε ασυμμετρίε και αυθαιρεσίε στην εφαρμογή του. Ο νόμος αυτό του 1988 εφαρμόζεται με αναδρομική ισχύ. Αυτό είναι ένα πρώτο πρόβλημα που είναι προφανέ. Και θα ήθελα να μάθω εδώ τη γνώμη των εκπροσώπων της Ισπανικής κυβέρνησης ό,τι αφορά την αναδρομική ισχύ αυτού του νόμου περί οκτών. Είναι ασύμετρη αυτή η εφαρμογή και πολύ ιδιόρυθμη και ιδιότροπη, γιατί παραδοσιακοί οικισμοί όπως είναι ο οικισμός ψαράδων του Τσοβίτο στην Τενερίφε, για παράδειγμα, ε, κατεδαφίστηκε ουσιαστικά ολόκληρος οικισμός παραδοσιακός και μάλιστα άρων-άρων, ενώ τεράστια ξενοδοχειακά, ξενοδοχειακά συγκροτήματα μένουν άθικτα. Πολύ ύποπτη είναι αυτή η διακριτική εφαρμογή του νόμου. Φαίνεται ότι εδώ πριτάνευσαν τα συμφέροντα τεράστιων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων έναντι των ε, νόμιμων ε, συμφερόντων, παραδοσιακών οικισμών, οικισμών ψαράδων ή άλλων παραδοσιακών οικισμών που έχασαν τα δικαιώματά τους εν μία νυχτή. Αυτές τις ασυμμετρίες στην εφαρμογή του νόμου θα πρέπει να τις εφαρμόσουμε. Δεν μπορεί να εφαρμόζεται με καπρίσιο αυτός ο νόμος. Δεν θα πρέπει να είναι διαφορετική η μεταχείριση ανάλογα με το σε ποιον ανήκει το κτίσμα, αν είναι μεγάλο ξενοδοχείο, αν είναι μικρό, μικρό σπίτι. Η συμφωνία του Άρχους που μας επισήμανε η κυρία Άουγκεν απαιτεί, και περιλαμβάνεται στο κοινοτικό κεκτημένο, απαιτεί μία πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία και στην ενημέρωση. Από ό,τι ξέρω, κάποιοι ιδιοκτήτε πήγαν στο αρχείο κινήτων και μέσα σε μία μέρα έμαθαν ότι έχασαν τα δικαιώματά τους. Μέσα σε μία μέρα έχασαν τα δικαιώματά τους. Υπήρξε μία διαδικασία που σίγουρα παραβίασε την συνθήκη του άρχους. Θα πρέπει λοιπόν να απαιτήσουμε η διοικητική, η διαδικασία να μην ε, παρακάμπτει την υποχρέωση συμμετοχής ή πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. Επίσης, σε ό,τι αφορά την απώλεια του δικαιώματος κυριότητας, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο που θα πρέπει να το προσέξει η Ισπανική κυβέρνηση. Και εκεί να εξεταστούν ίσως μετεγκαταστάσεις κάποιων οικισμών, γιατί μερικές φορές ε, οι πολίτες χάνουν και το μοναδικό του σπίτι, το οποίο έκτισαν με κόπους ε, μια ζωής και βρίσκονται από τη μία στιγμή στην άλλη χωρίς καμία εναλλακτική λύση. Υπάρχει αυτό το θέμα των μετακαταστάσεων πιθανών και υπάρχει και το θέμα των αποζημιώσεων που είναι υποχρεωτικό. Ένας άνθρωπος που έχει ένα σπίτι σε οποιαδήποτε παράκτια περιοχή και, τη, και το χάνει από τη μια στιγμή στην άλλη και μάλιστα χωρίς να λαμβάνει αποζημίωση, αυτό παραβιάζει όχι μόνο το κοινοτικό δίκαιο και το ισπανικό δίκαιο, αλλά και στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα επίσης η ισπανική διοίκηση και η ισπανική κυβέρνηση να δώσει απάντηση ατομικά σε κάθε τούντα σε κάθε υποβάλλοντα αναφορά. Αύριο θα ακούσουμε τους ε, αναφερόμενους και θα πρέπει να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση και με τη δική μας βοήθεια να δώσει απάντηση σε κάθε αναφορά με σεβασμό του κοινοτικού κεκτημένου αλλά και της εθνικής νομοθεσίας. Εγώ δεν συμφωνώ ότι με αυτό το πρόσχημα θα πρέπει να διώξουμε την Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή υπό αυτό το κριτήριο θα μπορούσε τώρα να μπει η Ισπανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό είναι μια υπερβολική δήλωση. Αλλά θα πρέπει εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ικανοποιήσουμε όλου του ετούντε. Γιατί όλε οι αναφορέ είναι είναι και θα πρέπει να σταθούμε στο ύψο των περιστάσεων και να συνεργαστούμε με την Ισπανική διοίκηση και την Ισπανική κυβέρνηση για να βρούμε μια λύση για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν ευσταθούν όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα για την Ισπανική κυβέρνηση και τον νόμο περιακτών, ισχύουν πολύ περισσότερο για ένα νησί της Ισπανίας, τη Φορμεντέρα που έχει έκταση 79 ε, τετραγωνικά χιλιόμετρα ε, και μέσα, στο μέσα στη χρονιά ζουν 5.000 άνθρωποι, 35.000 το καλοκαίρι. Πρόκειται για ένα νησί δηλαδή με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Πριν από λίγα χρόνια ήταν ένα πολύ φτωχό νησί, σχεδόν ακατοίκητο και οι κάτοικοι της Φορμεντέρας έγιναν εργολάβοι που έχτισαν με τα χέρια τους ε, τους πρώτους τουριστικούς οικισμούς και τα πρώτα εστιατόρια, ζουν ουσιαστικά από τον τουρισμό και αποτελούν υπόδειγμα πολεοδομίας φιλικής προς το περιβάλλον και υπόδειγμα κατασκευής με σεβασμό του περιβάλλοντος και της ιδιαιτερότητας του νησιού. Ουσιαστικά ήταν οικογενειακές οι επιχειρήσεις ε, που άρχισαν να λειτουργούν πριν από 40 χρόνια στο νησί. Το ξενοδοχείο Ροκαμπέγη ήταν το πρώτο ξενοδοχείο που χτίστηκε στη Φορμεντέρα ή το εστιατόριο Blue Bar που απέκτησε διεθνή φήμη και χρησιμοποιήθηκε για να διαφημιστεί και να προωθηθεί και στο εξωτερικό η φήμη αυτού του νησιού. Αν γνωρίζετε τη Φορμεντέρα θα ξέρετε το εστιατόριο Μόλι Ντεσάλικα ως Μινίστρα. Όλα αυτά τα, τα κτίρια είναι νόμιμα και μάλιστα έχουν μία ιστορία και μία αξία που είναι γνωστά στο νησί και μάλιστα κατασκευάστηκαν νόμιμα και με υλικά πολύ φιλικά προς το περιβάλλον. Μάλιστα μεταξύ κάθε κτίσματος υπάρχουν 150 μέτρα. Τα τελευταία 40 χρόνια δεν έχει αναγερθεί κανένα νέο κτίριο. Νομίζω είναι υπόδειγμα προστασίας του περιβάλλοντος η Φορμεντέρα και σήμερα με τον νόμο περιακτών το νησί αυτό θα χάσει την ταυτότητά του, θα χάσει το τη βασική πηγή πλούτου του που είναι ο τουρισμός και θα χάσει ουσιαστικά το σήμα κατά τεθέν. Γιατί οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων και των εστιατορίων θα χάσουν τις περιουσίες τους εξαιτία αυτής της εκχώρησης που θα γίνει στο κράτος. Και μάλιστα στερούνται οποιοδήποτε ενδικού μέσου γιατί δεν μπορούν ούτε να υποθηκεύσουν την περιουσία τους, δεν μπορούν να την μεταβιβάσουν, να την μεταγράψουν, γιατί δεν έχουν τέτοια δικαίωμα πια, έχουν μόνο δικαίωμα χρήσης. Έτσι δεν θα μπορέσουν να φροντίσουν όλες αυτές τις εγκαταστάσεις που είναι το χαρακτηριστικό της Φορμεντέρας. Και πολλοί φοβούνται στο νησί ότι θα αμεληθεί το νησί, θα μεληθούν όλες αυτές οι εγκαταστάσεις, μια οι ιδιοκτήτες του που θα πάψουν πια να είναι ιδιοκτήτες δεν θα ενδιαφέρονται να ανακαινήσουν και να συντηρούν αυτά τα κτίρια. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα κτίσματα βρίσκονται σε κατάφυτες περιοχές και μάλιστα η, ήδη η περιφερειακή αυτοδιοίκηση της Φορμεντέρα απαγορεύει το κτίσιμο σε πιο κοντά από 350 μέτρα από την ακτή και έτσι προστατεύεται και το περιβάλλον και το τοπίο στη Φορμεντέρα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ισπανική κυβέρνηση που ασκεί και την Προεδρία αυτό το εξάμεινο τα εξή. Καταρχήν, όλοι οι θύνοντες της Ισπανικής κυβέρνησης ε, ανέλαβαν τη δέσμευση για ένα ειδικό σχέδιο για τη Φορμεντέρα και μια δίκαιη οριοθέτηση για το νησί αυτό. Και μάλιστα η Μαρία Τερέσα Φράγκη Δελαβέχα, η αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, μαζί με πολλού υπουργού, επισκέφθηκα το νησί τα τελευταία χρόνια, αλλά δυστυχώ καμία πρόταση δεν έγινε. Πότε θα υποβληθεί το ειδικό σχέδιο για τη Φορμεντέρα για να ησυχάσουν επιπλέον οι κάτι, επιτέλου οι κάτοικοι αυτού του νησιού. Δικαίωμα, δίκαιο και δημοκρατία σημαίνει νομική ασφάλεια, ασφάλεια δικαίου. Σαφεί κανόνε χρειαζόμαστε για να ξέρουμε τι θα συμβεί σήμερα και τι θα συμβεί αύριο. Ο νόμος περί ακτών δυστυχώς ε, δεν εξασφαλίζει αυτή την ασφάλεια δικαίου και καταστρατηγεί τη δημοκρατία. Το πρόβλημα δεν είναι ο ίδιος ο νόμος. Ο νόμος περί είναι σωστός. Η εφαρμογή του είναι αλατωματική. Σε ό,τι αφορά την αναδρομική ισχύ. Είναι πολύ προβληματικό αυτό το ζήτημα της αναδρομικής αρχής, ιδιαίτερα όταν παραβιάζει το δικαίωμα κυριότητας. Ο νόμος σχεδιάστηκε για καταστάσεις που είναι τελείως άσχετες με την πραγματικότητα της Φορμεντέρας και με την κατάσταση πολλών από τους αναφερόμενους που διεκδίκησαν τα τελευταία χρόνια τα δικαιώματά τους, αλλά ματέως. Εμείς ζητούμε μια δίκαιη οριοθέτηση για τη Φορμεντέρα το σεβασμό τη ε, ιδιωτική ιδιοκτησία, την περιπτωσιολογική ανάλυση, την κατάργηση της αναδρομική ισχύω και ιδιαίτερα ε, ένα ειδικό καθεστώς για τη Φορμεντέρα. Και μάλιστα η παραχώρηση 60 ετών, μια και έχει περάσει ήδη τα 20, έχουν ήδη περάσει τα 20 χρόνια, δημιουργεί προβλήματα στη Φορμεντέρα, προβλήματα επιβίωση για το μέλλον αυτοί που έχτισαν πριν από 40 χρόνια έχτισαν μικρέ επιχειρήσει. Αυτοί θα την πληρώσουν. Ενώ τα μεγάλα ξενοδοχεία που χτίστηκαν πολύ αργότερα δεν χτίστηκαν στην παραλία, στι ακτέ. Αυτά τα τεράστια ξενοδοχεία είναι που ε, αλλοιώνουν το τοπίο του νησιού, αλλά αυτά τα ξενοδοχεία δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Δεν θα κυνηγήσει κανένα αυτούς, αλλά θα κυνηγήσει του ε, ιδιοκτήτε των μικρών επιχειρήσεων. Αυτό έχει εξοργήσει όλα τα συνδικάτα, όλα τα κόμματα στη Φορμεντέρα. Έχει δημιουργήσει ένα κίνημα. Υπήρξε υπόσχεση από την κυβέρνηση για ένα ειδικό καθεστώ για τη Φορμεντέρα, αλλά μέχρι στιγμή μόνο λόγια ακούσαμε και καμία έμπρακτη ε, δέσμευση πρόταση. Πότε επιτέλου θα υποβληθεί από την Ισπανική κυβέρνηση το ειδικό καθεστώ και σχέδιο για τη Φορμεντέρα. Ευχαριστώ. Κύριο Μαρτίνε. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της πενικής Κυβέρνησης που με πολύ συνοπτικό αλλά εμπεριστατωμένο και σαφή τρόπο μας εξήγησαν τον τρόπο εφαρμογής του νόμου περιακτών και γυαλού. Και μάλιστα μερικοί συνάδελφοι είπαν ότι ο νόμος περί ο καθεαυτός είναι καλός, άλλον δεν εφαρμόζεται σωστά. Πάντως ε, προβλέπει κάποιους, κάποιες βασικές αρχές αυτός ο νόμος. Αλλά ή θα είναι καλός ο νόμος και στην εφαρμογή του ή θα είναι κακός. Δεν μπορεί να λέμε ότι ο νόμος είναι καλός αλλά η εφαρμογή του είναι κακή. Γιατί στην εφαρμογή εφαρμόζονται κάποια θεμελιώδη στοιχεία του νόμου. Εγώ πιστεύω ότι και ο νόμος περί ακτών είναι καλός αλλά και σωστά εφαρμόζεται. Απλώς επειδή είναι περίπλοκος είναι λογικό να αντιμετωπίζει και προβλήματα στην εφαρμογή του, γιατί η κατάσταση είναι περίπλοκη και η εφαρμογή το ίδιο. Θα ήθελα να εμείνω σε κάτι που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να αγνοούμε ή να απαξιώνουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε απλούστατα ότι δεν μπορεί να, χαρακτηρίσει, να διαπιστώσει καταστρατήγηση της κοινοτική απλουστατα οτι δεν μπορει να χαρακτηρισει να διαπιστωσει καταστρατηγηση της κοινωτικη νομοθεσιας Και μάλιστα δεν το είπε μία φορά μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το είπε και το ξαναείπε. Δεν υπάρχει εδώ περίπτωση καταστρατήγησης του κοινοτικού δικαίου. Μιλούμε λοιπόν για παραβιάσεις εικαζόμενες, υποτιθέμενες, που μπορεί να μας αγγίζουν ή να μας συγκινούν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία. Αναφέρθηκε επίσης κάτι πολύ σημαντικό από την Επιτροπή. Το πρωτόκολλο που στηρίζεται στη συνθήκη της Βαρκελόνης. Κανένας δεν έλαβε υπόψη αυτό το σχόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το πρωτόκολλο όμως είναι ένα πρωτόκολλο που ευθυγραμμίζεται σε όλα τα σημεία με το περιεχόμενο του νόμου περιακτών και γυαλού. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το έγγραφο είναι πρωτοποριακό και παράδειγμα προς και για τους υπόλοιπους που θα εφαρμόσουν αυτό το πρωτόκολλο και θα το εφαρμόσουν σε κάθε εθνική νομοθεσία. Έχουμε λοιπόν το πρωτόκολλο που έχει υποδειγματική αξία που θα είναι ορόσημο και για πολλές χώρες θα αποτελέσει τον ακολουθηταίο κανόνα. Και αυτός ο κανόνας εφαρμόστηκε και στο νόμο περιακτών της Ισπανικής κυβέρνησης. Άκουσα ορισμένα σχόλια που πραγματικά με εξέπληξαν. Με εξέπληξε για παράδειγμα το γεγονός ότι πολλοί φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνω ότι το προσωπικό συμφέρον θα πρέπει να είναι υποδέστερο του γενικού συμφέροντος. Γιατί μερικοί στην ε, εξαιτία της ιδεολογίας της πολιτικής σου παράταξης θεωρούν την, το ιδιωτικό συμφέρον υπέρτερο αγαθό που υπερισχύει του συλλογικού συμφέροντος. Δεν είναι όμως αυτό βασική αρχή που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γενικό συμφέρον είναι αυτό που υπερισχύει του ιδιωτικού συμφέροντος ορισμένων ομάδων, λίγων. Ενώ το αντίθετο άκουσα. Ορισμένοι εδώ διατρανώνουν ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία, η ιδιωτική περιουσία είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Δηλαδή θα πρέπει να ε, διευρύνουμε τη διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το δικαίωμα της ε, ιδιωτικής περιουσίας. Θα σηκωθεί από τον τάφο του ο Είναι, είναι ανθρώπινο δικαίωμα η ιδιωτική περιουσία, αν είναι δυνατόν. Θα πρέπει τότε στη συνθήκη των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων να δούμε αν όντως η ιδιωτική περιουσία αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Και άκουσα και ένα άλλο σχόλιο που με ανησύχησε, που μπορεί να έχει κάποιο δίκιο. Άκουσε λοιπόν ότι όταν κάποιος είναι ιδιοκτήτης μιας εγκατάστασης, με μιας επιχείρησης, τη φροντίζει ως κόριο οφθαλμού, όταν όμως δεν είναι ιδιοκτήτης, αλλά έχει το δικαίωμα χρήση μόνο για 60-90 χρόνια, τότε ε, τα φορτώνει στον κόκορα και διαφορεί πλήρως για την επιχείρηση αυτή. Δηλαδή, το αν φροντίσει κάποιος ένα αγαθό ή μια επιχείρηση σχετίζεται με το κατά πόσο έχει δικαίωμα κυριότητα σε αυτό το αγαθό ή σε αυτή την επιχείρηση. Δεν λαμβάνει υπόψη ότι αυτή η επιχείρηση ε, του επιτρέπει να επιβιώσει αυτός και να συντηρηθεί η οικογένειά του. Το μόνο που ενδιαφέρει εδώ είναι ο τίτλος ιδιοκτησίας και όχι η επικαρπία, η χρήση και εκμετάλλευση αυτής της ιδιοκτησίας. Έτσι φαίνεται. Καθένα φροντίζει το αγαθό μόνο και μόνο, αν είναι ιδιοκτήτη. Αλλιώ αδιαφορεί πλήρω. Αυτό πραγματικά με προβλημάτισε. Θα ήθελα τώρα να πω κάτι προς τον κύριο Χέλμερ, που είπε κάποια στιγμή ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Είπε ότι το όνειρο πολλών Βρετανών είναι να περάσουν τη σύνταξή τους στις Ισπανικές ακτές. Ήταν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί οι Βρετανοί που είχαν όνειρο να περάσουν τη σύνταξή τους ε, στις Βρετανικές ακτές και εξακολουθούν να έχουν αυτό το όνειρο οι Βρετανοί συνταξιούχοι γιατί εκεί βρίσκονται στις Ισπανικές ακτές ε, απολαμβάνουν τα καλά μιας υπέροχης ηλιόλουσης χώρας και μιας φιλόξενης κοινωνίας, συμμετέχουν μάλιστα και στις περιφερειακές εκλογές και στις δημοτικές και στις εκλογές και δεν έχουν κανένα παράπονο, γιατί δεν έχουν κανένα λόγο να παραπονιούνται αυτοί οι Βρετανοί συνταξιούχοι. Και όταν είναι εκατομμύρια αυτοί που περνάνε ζωή και κότα στην Ισπανία, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση για τα συμφέροντα ελαχίστων που ναι μεν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, αλλά να θέσουμε τα πράγματα στο πλαίσιο τους και στο σωστό τους μέτρο και κλίμακα. Κύριε Έλμερ, με όλη την προπαγάνδα και τη διαφήμιση που κάνετε εσείς και άλλοι σαν και εσάς, που έχουν περιουσιακά στοιχεία, που έχουν ολόκληρες περιουσίες και που ε, αγοράζουν περιουσίες και σε άλλα σημεία και με την προπαγάνδα που κάνετε λέγοντας ότι εγώ δεν θα συμβούλευα κανένα ψηφοφόρο μου να πάει και να αγοράσει στην Ισπανία. Πολύ πιθανό κάποιος φίλος του κύριου Έλμερ έχει συμφέροντα σε άλλες ε, ευρωπαϊκές χώρες και σε άλλες ακτές. Εκεί ίσως θα συμβουλεύετε τους ψηφοφόρους σας να αγοράζουν σε άλλες χώρες και σε άλλες περιοχές. Διαδικαστικό. Διαδικαστικό παρακαλώ να παραφέρετε στην τάξη τον κύριο Μαρτίνες, κύριε Πρόεδρε. Μια στιγμή, μια στιγμή. Συνάδελφοι Μαρτίνες, κύριε Πρόεδρε, ζητώ το δικαίωμα να απαντήσω, Πρόεδρος. Θα τελειώσει ο συνάδελφος και μετά θα απαντήσετε αν χρειάζεται. Εγώ δεν είπα. Ε, μακρηγορήσατε κύριε Μαρτίνες, παρακαλώ ολοκληρώστε. Είπα ότι ο κύριος Έλμερ δήλωσε ότι θα συμβούλευε τους ψηφοφόρους του να μην αγοράσουν σπίτι στην Ισπανία. Αυτό είπα. Ο ίδιος ο κύριος Έλμερ το δήλωσε αυτό. Το είπατε κατά λέξη κύριε Έλμερ, αυτό είπατε. Εγώ δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο στους Βρετανούς. Εγώ θα έλεγα στους ψηφοφόρους του κ. Έλμερ να έρθουν και να ε, μιμηθούν τους εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες τους που αγόρασαν στην Ισπανία και περνάνε μια χαρά στα σπίτια που αγόρασαν στην Ισπανία. Και πραγματικά είναι τεράστια τα συμφέροντα αυτού του κλάδου. Και μερικές φορές τα συμφέροντα αυτού του κλάδου έχουν ε, ακριβώς επειδή έχουν συμφέροντα σε άλλες περιοχές και σε άλλες ε, ακτές και σε άλλες χώρες, κάνουν προπαγάνδα εις βάρος της Ισπανίας. Και ακριβώς οι ισπανικές ακτές, εξαιτία ε, των καταχρήσεων που έγιναν στην αστικοποίηση, ε, υπέσαν τεράστιες ζημιές και ευτυχώς θεσπίστηκε ο νόμος περιακτών. Άλλωστε δεν είναι το ανώτατο Ισπανικό Δικαστήριο που έκρινε ότι είναι σωστή η αποζημίωση που προβλέπει την παραχώρηση για 60 χρόνια. Το συνταγματικό δικαστήριο το έκρινε, όχι το ανώτατο δικαστήριο. Το συνταγματικό Ισπανικό δικαστήριο θεώρησε σωστή μία αποζημίωση που αντί για την ε, κυριότητα προβαίνει σε 60 ετή επικαρπία. Το Συνταγματικό Δικαστήριο θεωρεί ότι επικαρπία για 60 χρόνια μίας περιουσίας είναι μια δίκαιη αποζημίωση για κάποιον που χάνει την κυριότητα ενός ακίνητου. Και σε τέτοια περίπτωση ε, εφαρμόζεται ο νόμος περιακτών και η ιδιωτική περιουσία, ένα συγκεκριμένο ακίνητο, περνάει στη δημόσια περιουσία με αυτή την αποζημίωση που είναι η επικαρπία για 60 χρόνια. Αυτά και ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις που είχα, που είχα σημειώσει. είσαι, Στέρα. are you going to give my colleague, Mr. Helmer, the right to reply to this outrageous suggestion from Mr. Martinez Martinez before I make my contribution? Collega, un minuto però.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 Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Μαρτίνες ε, είπε ότι αναφέρθηκα σε εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπων που έχασαν τα σπιτία του, Όχι, εγώ είπα δεκάδες. Ε, ε, είπε ότι κάποιοι είναι ικανοποιημένοι. Ε, ναι, ε, σε πολλούς επιτίθενται άνθρωποι στον δρόμο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε με αυτούς. Ε, με πολύ άσχημο τρόπο έχει απαλωτριωθεί πολλών ανθρώπων τα κίνητα έχουν απαλωτριωθεί στην η Ισπανία. Ε, και επίση ο κύριος Μαρτίνε υπονόησε ότι έχω προσωπικό συμφέρον. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και επίση είπε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα και σε άλλε χώρε ε, ε, στη Μεσόγειο. Θα πρέπει να πω ότι κατά τη διάρκεια των ετών έχω λάβει αναφορέ παράπονα και από άλλε χώρε, αλλά το 90% αφορούσαν την Ισπανία και δεν αφορούσαν άλλε χώρε. Ο κύριος Τσίσεστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να επανέλθω στο βασικό θέμα της συζήτησης. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους την, ε, το, το παλιό ρητό ότι ο δρόμος για την κόλαση ε, είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Και νομίζω ότι πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Ο νόμος αυτός έχει καλούς, καλές προθέσεις, έχει όμως κακά αποτελέσματα. Μέχρι την παρέμβαση του κυρίου Μαρτίνες, είχα εκπλαγεί θετικά από τον αριθμό συναδέρφων από την Ισπανία που μίλησαν για τις αδικίες προς ε, μεμονωμένα άτομα ε, όσον αφορά την περιουσία τους στην υπόθεση αυτή. Ξέρω ότι ο κύριος Μαρτίνες ε, απολαμβάνει που δίνει ζωή στη συζήτηση, εντάξει, αλλά θα πρέπει να απαντήσω με ανάλογο τρόπο στον κύριο Χέλμερ ότι ε, ε, με ανάλογο τρόπο με τον κύριο Χέλμερ ότι και εγώ έχω λάβει πολλές επιστολές σχετικά με θέματα ακινήτων στην Ισπανία και εμένα οι συμβουλές μου θα ήταν οι ίδιες για να αποφύγουμε τον κίνδυνο εμφάνιση τέτοιου προβλήματο. Θα, θα έλεγα δηλαδή στον κόσμο να μην αγοράσει ακίνητα στην Ισπανία. Δυστυχώ όμω, ε, πολλοί κόσμοι δεν, άκουσε, δεν εισάκουσε τι ε, συμβουλέ αυτέ. Ε, αγόρασαν ακίνητα και έχουν συναντήσει δυσκολίε. Προφανέ σήμερα είναι ότι εμεί που ανησυχούμε σχετικά με τους μα μας από τι χώρε μα όσον αφορά τα δικαιώματα κινήτων τους στην Ισπανία. Σε αυτούς προστίθενται και πάρα πολλοί Ισπανοί υπήκοοι και εμένα με εκπλήσει το πώ η Ισπανία μπορεί να φέρεται έξω στους δικούς της υπηκόου. Ε, δεν, δεν υπάρχουν σωστές διαδικασίες, δεν υπάρχει αποζημίωση, ε, αυθαίρετη ε, κατάσχεση ακινήτων. Ε, αυτό είναι σαν ε, απολυταρχικό καθεστώς. Και σίγουρα δεν είναι κάτι τέτοιο η Ισπανία. Θα ήθελα πολύ να δω να αλλάζει η κατάσταση. Θα ήθελα να επενέσω τους εκπροσώπους της ε, Ισπανικής ε, κυβέρνησης για το θάρρος τους που ήρθαν εδώ πέρα και ελπίζω να μεταφέρουν το μήνυμα σημαντικής ανησυχίας, ε, οργής που νιώθει ο κόσμος για την κατάσταση αυτή και να κάνουν κάτι για να διορθώσουν την κατάσταση. Και η τελευταία μου παρατήρηση, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι θυμάμαι στις ακτές της ε, Βόρειας Ισπανία στον δρόμο προς το Σανταντέρ το 1982, που παρατήρησα, πριν πολλά χρόνια δηλαδή, μεγάλο όγκο ε, παράκτιας ανάπτυξης ε, και αναρωτήθηκα. Γιατί έχει επιτραπεί η περαιτέρω ανάπτυξη των περιοχών. Γιατί έχουν επιτρέψει οι αρχές κάτι τέτοιο τη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος και γιατί επιτρέπεται σε πολλούς, σε πολλά αθώα θύματα να χάνουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους, χωρίς να λαμβάνουν αποζημίωση. Συγγνώμη, αλλά αυτό δίνει πολύ κακό όνομα στην Ισπανία. Δεν σας βοηθάει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν συνεχίζετε το σκάνδαλο αυτό και σας καλώ να κάνετε κάτι για να διορθώσετε την κατάσταση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Βόλης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω τον πρόσωπο της ισπανική κυβέρνηση Σίγουρα δεν ήταν εύκολο για αυτό να έρθει εδώ σήμερα. Οι εξηγήσει σα όσον αφορά τον νόμο ε, είναι χρήσιμε. Θα ήθελα να πω ότι οι στόχοι σίγουρα είναι ευγενείς, ε, θα πρέπει να τους επενέσουμε και ε, μου θυμίζουν την περιοχή, την παράκτια περιοχή που εκπροσωπώ εγώ στο Ανατολικό Γιόξια, όπου έχουμε παρόμοια πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όχι το θέμα της ε, οικοδόμησης των ακτών, αλλά το θέμα της διάβρωσης των ακτών και θα πρέπει να βρούμε τρόπο διαχείρισης των ακτών και να ε, βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που μπορεί να χάσουν τα σπίτια τους. Αυτό όμως ε, είναι αποτέλεσμα κάποιου φυσικού φαινομένου. Αυτό που γίνεται εδώ πέρα όμως είναι πράξη των κυβερνήσεων και των αρχών. Και ο τρόπος εφαρμογής του νόμου φαίνεται να δημιουργεί το πρόβλημα και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυσανάλογα επηρεάζει ε, Ευρωπαίους πολίτες που παρέχονται από άλλα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Δεν θα είχαμε τέτοιο αριθμό αναφορών στο τραπέζι μας εάν δεν υπήρχε πραγματικό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις αναφορές αυτές. κατά κάποιο τρόπο με ενοχλεί περισσότερο η αντίδραση της Κομισιόν, διότι για μένα πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχουμε ενθαρρύνει τον κόσμο και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου να ε, επωφεληθούν από το δικαίωμα ελεύθερη κινητικότητα σε όλη μας την Ήπειρο. Και συμφωνώ με τον κύριο Μαρτίνες ότι Πολλοί άνθρωποι το κάναν αυτό χωρίς προβλήματα, χωρίς δυσκολίες. Είναι σαφές όμως από την ιστορία του φακέλου αυτού στην Επιτροπή μας κατά τη διάρκεια των ετών ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ανθρώπων από διάφορα κράτη-μέλη της, Ευρώπη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήγαν στην Ισπανία και συνάντησαν σημαντικά προβλήματα, έχασαν περιουσίες, έχασαν ε, τα κίνητά τους και αυτό ε, θα πρέπει ε, να αποτελεί αντικείμενο αποζημίωσης. Εάν η ε, Ευρώπη δεν μπορεί να βοηθήσει εγώ ως υποστηρικτής της Ευρώπης θα απογοητευτώ πάρα πολύ διότι πιστεύω ότι έχουμε ευθύνη τη στιγμή που ενθαρρύναμε την ελεύθερη κινητικότητα να διασφαλίσουμε ένα δίκαιο σύστημα σε όλη την Ευρώπη για τους πολίτες μας, το οποίο να αξίζει το όνομά του. Και εάν δεν παρεξήγησα το περιεχόμενο, ακριβώς αυτό αναφέρεται στο πρόσφατο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Ισπανικής Κυβέρνησης. Φαντάζομαι δεν είναι και πολύ εύκολη θέση της. Θα ήθελα να αναφερθώ σε πολλά που ακούσαμε σήμερα, για παράδειγμα αυτά που είπε ο κύριο Μάτο. Το δικαίωμα τη ιδιοκτησία είναι βασική αρχή τη κοινωνία μα. και μία παραβίαση του δικαιώματο αυτού δημιουργεί μία έλλειψη ασφάλεια δικαίου. Ο κύριος Μέλμερ είπε ότι θα συμβούλευε κανέναν εκλογέα να αγοράσει περιουσία ή σπίτι στην Ισπανία. Επίση, αυτά που ακούσαμε από την κυρία Στάρα για τη Φορμεντέρα είναι συγκλονιστικά. Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις της Και είμαι σίγουρη, σίγουρος ότι αύριο που θα ακούσουμε τους ετούντες ε, για τις περιπτώσεις τους να αντιληφθούμε και άλλες τέτοιες καταστάσεις. Σίγουρα είναι προβληματική η εφαρμογή του νόμου περί ακτών, όπως φάνηκε από αυτά που ακούσαμε σήμερα. Και όχι μόνο είναι προβληματική η εφαρμογή του νόμου, αλλά ο ίδιος ο νόμος δεν είναι τόσο καλός όσο πιστεύαμε στην αρχή. Και μάλιστα η αναδρομική ισχύς ε, του νόμου αυτού έχει ολέθριο αποτέλεσμα για χιλιάδες οικογένειες. Ερωτώ λοιπόν για την αποζημίωση για την απώλεια ιδιοκτησίας, για την απώλεια περιουσίας. Αναφέρθηκε το θέμα της αποζημίωσης, αλλά όχι επαρκώς κατά τη γνώμη μου. Ο νόμος πυριακτών θεσπίζει ως δικαίωμα αποζημίωσης την παραχώρηση της χρήσης ως αποζημίωση για το απώλεια του δικαιώματος κυριότητας. Φαίνεται ότι ούτε αυτές τις παραχωρήσεις χρήσης κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν προβλέπεται αυτεπάγγελτη παραχώρηση από την ε, Ισπανική ε, Αρχή, αλλά υποβολή προηγούμενης αίτησης από τους θυγόμενους. Και μάλιστα η εκπρόσωπος Τη ισπανική κυβέρνηση είπε ότι στηρίζεται στο νόμο πειρακτών για να διορθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά τι προβλέπει να κάνει η κυβέρνηση για να αποκαταστήσει μια ασφάλεια δικαίου που έχει διαταραχθεί με την εφαρμογή αυτού του νόμου. Επίσης, το κριτήριο της παροχής ε, ε, παραχώρησης ε, δεν θα το συνοδεύσετε από καμία χρηματική αποζημίωση. Παρόλο που ο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων προβλέπει το δικαίωμα δίκαιη αποζημίωση και την απαλωτρίωση. Ευχαριστώ, κύριε Χιμένες. Ως Ισπανίδα δεν ε, αισθάνομαι και ιδιαίτερη εφορία με τη συμμετοχή μου σε αυτή τη συζήτηση και μάλιστα η δυσαρέσκειά μου οφείλεται σε δύο λόγου. Καταρχήν στις επικρίσεις που ακούεις βάρος της χώρας μου που πραγματικά με πονάμε πολύ, αλλά συγκινούμε και από την παρουσία των θυμάτων που μερικές φορές με δάκρυα στα μάτια μας εξιστορούν ε, την κατάστασή τους. Μάλιστα είμαι και μέλος της ε, Επιτροπής Πολιτικών ε, Ελευθεριών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχω λάβει πολλές αναφορές και πολλά mail με προβλήματα και καταστάσεις από πολλές χώρες. Δεν μπορώ να μένω λοιπόν αδιάφορη γιατί εγώ περνάω ε, τα καλοκαίρια μου στην Ανταλουσία και μάλιστα από την ίδια την πατρίδα μου ε, λαμβάνω επιστολές απελπισμένων συμπολιτών μου που λένε θα χάσουμε τα σπίτια μας από το νόμο αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιος τρόπος να εφαρμόζουμε ένα τέτοιο νόμο. Υπάρχει τεράστια κοινωνική κατακραυγή για την εφαρμογή αυτού του νόμου. Εγώ από μικρή έμαθα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και γι' αυτό έγινε και βουλευτής. Τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να τάσσονται υπέρ της αξιοπρέπειας και της δικαιοσύνης ε, προς τα θύματα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ε, προστατεύουμε τα θύματα και την ε, δικαιοσύνη και την αξιοπρέπειά τους. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ακούσουμε τους θυγόμενους, θα πρέπει να τους ξαναδώσουμε τη σωστή τους θέση. Αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα. Έχω και κάποιες τεχνικές ερωτήσεις που θα μπορούσα να τις κάνω και τώρα, αλλά προτιμώ να ακούσουμε αύριο τους υποβάλλοντες στην αναφορά. Θα ήθελα να ρωτήσω πραγματικά αν ε, συμπεριφέρεστε δίκαια προς αυτούς τους ανθρώπους. Αν μου πάρετε το σπίτι μου, θα πρέπει να λάβω μια δίκαιη αποζημίωση. Τι θα πει όμως δίκαιη αποζημίωση, πώς ε, αποτιμάτε εσείς τη δίκαιη αποζημίωση. Γιατί είπατε ότι για τι απαλωτριώσει θα δώσετε αποζημίωση. Ποια είναι για εσά η δίκαιη αποζημίωση, Γιατί επαναλαμβάνω, έχει ξεσηκωθεί ο κόσμο, έχει δημιουργηθεί τεράστια κατακραυγή, γιατί πολλοί χαρακτηρίζουν άδικε αυτέ τι αποζημιώσει. Σα ευχαριστώ. Κολέγα Άντερσεν. Άντερσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ εκπροσωπώ τους Βρετανούς της Νότιας Αγγλίας. Και το κάνω αυτό γιατί ήρθαν πάρα πολλοί Βρετανοί και μου είπαν ότι χάνουν τα σπίτια τους. Αλλά είμαι και Ισπανός, Ισπανίδα επίκος ταυτόχρονα. Γι' αυτό προβληματίζομαι πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει στη χώρα μου. Επισκέφτηκα επιτόπια ορισμένα σημεία που είχαμε τέτοια κρούσματα και ερεύνησα και κατέληξα στο συμπέρασμα, δεν θα το πιστεύετε, αλλά τα 80% των ανθρώπων που πέστησαν αυτή τη ζημιά είναι οι Ισπανοί. Κύριε Μαρτίνες, μιλάμε για 400.000 οικογένειες που τις αφορά το πρόβλημα αυτό. Δεν μπορείτε εύκολα να πείτε «Α, είναι ασήμαντο». ζήτησε από το Κοινοβούλιο συζήτηση και ψήφισμα. Κατ' επανάληψη, γιατί το πρόβλημα αυτό χρονίζει. Χρονίζει στην Επιτροπή μας. Λύση δεν έχει δοθεί. Και όσο πιο πολύ καθυστερούμε να λύσουμε το πρόβλημα, τόσο πιο πολύ θα χρειαστεί χρόνος για να λυθεί το πρόβλημα. Προστασία του περιβάλλοντος που είναι το κύριο πρόβλημα. Νομίζω οι περιφέρειες όπου συμβαίνουν αυτές οι ανομαλίες δεν θα πρέπει να ξαναπάρουν κοινωτικά κονδύλια. Γιατί είτε ο νόμος του Ιγιαλού είναι θέμα της Ένωσης ή όχι, το θέμα είναι ότι αυτές οι ανομαλίες και τα βάσανα όλων αυτών των ανθρώπων, ασχέτως εθνικότητας, δεν μπορεί να εξακολουθούν να συμβαίνουν όπως γίνεται. Η Ένωση δεν μπορεί να εξακολουθεί να χρηματοδοτεί αυτές τις περιοχές. Και έχω και μερικές ερωτήσεις προς την πρόσωπο του Υπουργείου. Γιατί η κυβέρνηση στερεί όλους τους ανθρώπους αυτούς από τα σπίτια τους με βάση αυτό το νόμο περί ακτών Αιγιαλού, αλλά τους ζητάει να πληρώνουν, να ξεπληρώσουν τις υποθήκες και τα χρέη που έχουν για τα σπίτια αυτά. It is often, it is often said. Συχνά ακούμε ότι το συνταγματικό δικαστήριο είπε ότι είναι συνταγματικός ο νόμος αυτός. Ή είπε όμως ότι η αναδρομική ισχύ του είναι συνταγματική. Κύριε Μαρτίνες, τρίτη ερώτηση προς την Ισπανική κυβέρνηση. Τι εγγυήσεις δίνει η Ισπανική κυβέρνηση σε κάποιον που θα θέλει να αγοράσει ένα σπίτι στην Ισπανία. Πρόεδρος. Και τελευταία συνάδελφος Γκουρμάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που ως γυναίκα πρόεδρος ε, μερικοί συνάδελφοι που chairman, chairman, τέλος πάντων. Βλέπετε πρέπει να πω είναι chairwoman. Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου ήρθε, μας μίλησε για το πρόβλημα αυτό. Πρέπει να βρούμε μια λύση και από ό,τι καταλάβαμε προτίθεστε να δώσετε μία λύση. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να σεβαστείτε και την εθνική σας νομοθεσία. Εγώ είμαι Ουγγαρέζα. Τα τελευταία τέσσερα καλοκαίρια πήγα στην Ισπανία. Το πρώτο αυτό δεν το, δεν το γνωρίζω. Ξέρω όμως, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Συνεχίζω στα Ουγγρικά. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μας είπε ότι οι επιμέρους περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων είναι πέραν των αρμοδιοτήτων της Κομισιόν. Τι είναι, είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα άθροισμα επιμέρους προβλημάτων. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να βρεθεί η λύση. Εγώ πιστεύω στην Ευρώπη και στην Ένωση Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να μάθουμε περισσότερο ο καθένα για τι άλλε χώρε, οι Βρετανού, οι Ούγγροι, οι Ολλανδοί, όποιο τέλο πάντων έχει αγοράσει περιουσία στην Ισπανία, θα πρέπει να γνωρίζει του όρου ε, κυριότητα και ιδιοκτησία στην Ισπανία και φυσικά πρέπει να σέβεται τον Ισπανικό νόμο. Οι αναφερόμενοι είναι παρόντες στην αίθουσα και περιμένουν ένα είδος νομικής αποκατάστασης. Θέλουν να γυρίσουν ε, στην πατρίδα τους αύριο το απόγευμα με μια λύση που να τους έχει προταθεί. Κατανοώ το ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση η Ισπανική κυβέρνηση, διότι το, η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι σαφής. Εμείς οι Ευρωβουλευτές δεν θέλουμε ο κόσμος να σταματήσει να αγοράζει σπίτια ή διαμερίσματα στην Ισπανία. Θέλουμε να πάνε στην ηλιόλου στην Ισπανία και να αγοράζουν κατοικίες. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί λύση. Πρέπει να προταθεί μια λύση στους αναφερόμενους. Και το μόνο που ήθελα να πω στους εκπροσώπους, στον εκπρόσωπο της Ισπανικής κυβέρνησης, που τη χαίρομαι που ήρθε εδώ, είναι η δουλειά της. Είναι η δουλειά τη γι' αυτό έχει εκλεγεί. Η Κομισιόν ενδεχομένως θα μπορούσε να μελετήσει λίγο πιο προσεκτικά το θέμα αυτό και να προτείνει μια λύση. Και πιστεύω ότι η Ισπανική κυβέρνηση στην περίπτωση αυτή θα συνεργαστεί. Πρόεδρος, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις σας. Είναι σαφές ότι η Επιτροπή μας θεωρεί ότι είναι της αρμοδιότητάς της το θέμα αυτό αυτών εδώ των αναφορών Νομίζω αυτή τη θέση την συμμερίζονται οι περισσότεροι σε αντίθεση με τη γνώμη της Κομισιόν. Σχεδόν ομόφωνα ε, οι συνάδελφοι έχουν μια συγκεκριμένη θέση για την Ισπανική νομοθεσία. και προσυπογράφουν τις καταγγελίες των αναφορών για υποτιθέμενες σοβαρές παραβιάσεις που αφορούν αρχές των συνθήκων και κοινωτική νομοθεσία που η Ισπανική κυβέρνηση δεν τηρεί αυστηρά. Θα ξαναδώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ισπανικής Κυβέρνησης με την ερώτηση που έκανε άμεσα ε, συνάδελφος Άριας Ετσεβαρίας. Τι σκοπεύει να κάνει η Ισπανική Κυβέρνηση. Η Επιτροπή Αναφορών αποφασίζει να δώσουμε συνέχεια και βάθος στο θέμα αυτό γιατί θεωρούμε πολύ σημαντικές τις αναφορές αυτές. Η Ισπανική κυβέρνηση τι σκοπεύει να κάνει. Αν έχετε κάτι να μας πείτε, πείτε το τώρα. Muchas Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν εδώ και μάλιστα μερικές φορές ήταν επανάληψη των ίδιων σημείων. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω μία σύνοψη και μία ανακεφαλαίωση. Καταρχήν διαπίστωσα ότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση και φάνηκε αυτό από τις παρεμβάσεις στην Επιτροπή σας. Γιατί ακούσαμε ότι θα χαθούν ε, κατοικίες και μάλιστα εν μία νυχτή. Και μάλιστα είπαν ότι αυτό συμβαίνει από το 2008. Και ο νόμος περιακτών που είναι από το 1988 δεν εφαρμόστηκε καθόλου μέχρι το 2008. Θα ήθελα να σας πω ότι ο νόμος περιακτών άρχισε να εφαρμόζεται από την αρχή. Και αυτό προσπάθησα να σας εξηγήσω με τις διαφάνειες που σας έδειξα. Από τη στιγμή που εγκρίθηκε, από το 1988 δηλαδή, άρχισε να εφαρμόζεται. Και μάλιστα το 1998 ήταν η χρονιά που οριοθετήθηκαν περισσότερα χιλιόμετρα ακτών. Το 1998. Τότε έγινε η μεγαλύτερη οριοθέτηση χιλιόμετρων για τα κατά πόσο ένα αγαθό ανήκει στην κρατική περιουσία ή όχι. Οπότε και το 1998 ιδιαίτερα που έγινε η μεγαλύτερη οριοθέτηση εφαρμόστηκε ένας νόμος που ήταν ενισχύ. Δεύτερη σύγχυση. Αναφέρθηκαν οι συνέπειες μιας οριοθέτησης ακόμη και για περιουσίες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ιδιωτικέ. Αναφέρθηκε η περίπτωση τη Εμπορία Μπράβα. Δεν έχει εγκριθεί ακόμη αυτή η οριοθέτηση, αλλά εκεί παραμένει η κυριότητα, η ιδιωτική κυριότητα στι περιουσίε αυτέ. Το μόνο που κρίνεται ω δημόσιο κτήμα είναι τα κανάλια, το νερό, που ούτω ή άλλω ήταν δημόσιο κτήμα και πριν την εφαρμογή του νόμου περιακτών το 88. Όλα αυτά τα σχόλια δημιουργούν κάποια σύγχυση. Φαίνεται ότι μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι και γίνονται ένα αχτάρμά πολύ διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ως προς το στόχο του νόμου περιακτών. Είναι να προστατευτεί μια πολύ ευάλωτη και πολύ στενή λωρίδα ακτών. Μερικές φορές ε, είναι λίγα δεκάδες, ε, μερικές δεκάδες μέτρα αυτή η ζώνη. Και στην ευάλωτη αυτή λεπτή λωρίδα πιστεύω ότι ε, το δημόσιο συμφέρον υπερισχύει του ιδιωτικού συμφέροντος. Ποια ήταν, ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του νόμου περιακτών που επικρίθηκε προσπαθήσαμε να ανακτήσουμε κάποιες θύνες, ζώνες με αμοθύνες που είχαν ε, πληγεί από την ανεξέλεγκτη οικοδόμηση. Προσπαθήσαμε να ανακτήσουμε κάποιους υγρότοπους, κάποιους βάλτους. Προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε το φυσικό περιβάλλον σε αυτές τις στενές ευαίσθητες λωρίδες των ακτών. Αυτό ήταν ο στόχος του νόμου περί ακτών που τόσο κατακρίθηκε. Και πρώτα απ' όλα θέλουμε να διαφυλάξουμε το περιβάλλον στην Ισπανία και τα δικαιώματα κυριότητας ιδιοκτησίας που μπορούν να μπορεί να έχουν μερικοί, τα μετατρέψαμε σε δικαιώματα εκχώρησης. Σε περίπτωση που τα κτίσματα ήταν νόμιμα, κάτι που δεν συμβαίνει για όλα τα κτίσματα, δεν πρόκειται να καταδεφιστούν. Τα νόμιμα κτίρια δεν πρόκειται να καταδεφιστούν και σίγουρα σε καμία περίπτωση άμεσα, αμέσως το δικαίωμα παραχώρησης ή εγχώρησης ισχύει για 60 χρόνια και μάλιστα το 1991 το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε συνταγματικό αυτό το νόμο περί ακτών. Και μάλιστα νομίζω ότι η κοινωνική λειτουργία αυτών των αγαθών και η περίσχυση του κοινωνικού τους ρόλου υπερισχύει του ιδιωτικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Και ακριβώς επειδή ορισμένες περιοχές ε, κρίθηκαν ως δημόσιο κτήμα, ως δημόσια περιουσία, έδωσαν ε, βάση για την απαλωτρίωση. Και μάλιστα ως αποζημίωση και καταρχήν γενικά προβλέφθηκε ότι ήταν δίκαιη και ισορροπημένη αυτή η παραχώρηση για 60 χρόνια. Ως αντικατάσταση του δικαιώματος κυριότητας που ε, απολέστηκε. Είμαστε δημοκρατική χώρα στην οποία ισχύει κράτος δικαίου, γι' αυτό και υποτασσόμαστε στην ομολογία του δικαστηρίου. Το συνταγματικό δικαστήριο έκρινε τη συνταγματικότητα αυτού του νόμου. Μπορεί να έχουν γίνει μεμονωμένα κάποιε καταχρηστικέ εφαρμογές, πάντως γενικώ η αποζημίωση που εφαρμόζουμε είναι η δίκαιη αποζημίωση. Τώρα για την οριοθέτηση που αναφέρθηκε ότι γίνεται αυθαίρετα, με αναδρομική ισχύ και ούτω καθεξής. Επαναλαμβάνω, η οριοθέτηση άρχισε να εγκρίνεται από το 88. Υπήρξαν οριοθετήσεις και πριν το 88. Γιατί δεν θέσπισε ο νόμος περί αυτό το, αυτή την αρχή του δημόσιου κτήματος στην Ισπανία και πριν το νόμο περί υπήρξαν κάποιες, κάποια αυθαίρετα επειδή ε, ήταν κατασκευές που έγιναν χωρίς πολλαδομική άδεια, είχαν γίνει σε περιοχές που είχαν ήδη χαρακτηριστεί ως δημόσιο κτήμα. Αυτός ο χαρακτηρισμός υπήρχε και πριν το 88. Αναφέρθηκε η περίπτωση του Τσοβίτο. Εκεί όλες, όλες, ε, όλες οι δίκες που έγιναν, όλες οι προσφυγές που κρίθηκαν στα δικαστήρια, έκριναν ότι όντως αυτές οι κατοικίες ήταν αυθαίρετες και είχαν οικοδομηθεί πάνω σε δημόσιο κτήμα. Άρα ήταν νόμιμη η απαλωτρίωση αυτών των οικισμών. Θα πρέπει να γίνει κάποια διάκριση, επαναλαμβάνω, μεταξύ παράνομων, οικισμών, ε, παράνομων κατασκευών και αυθαίρετων. Οι παράνομες ε, δεν έχουν κανένα δικαίωμα, ενώ οι νόμιμες έχουν αυτό το δικαίωμα της παραχώρησης για 60 χρόνια. Μάλιστα, έχει προβλεφθεί και δικαίωμα προσφυγής. Οι θυγόμενοι που έκριναν άδικη την ε, αποζημίωση, το χαρακτηρισμό, είχαν δικαίωμα άσκησης προσφυγής. Υπάρχει δικαίωμα καταρχήν διοικητική προσφυγής και επαναλαμβάνω, για τις οριοθετήσεις υπάρχει ένα, ένας πρώτος βαθμός στο πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο και σε δεύτερο βαθμό στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο. Στο ανώτατο δικαστήριο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα προσφυγής και στην πολιτική δικαιοσύνη. Και μάλιστα στις περισσότερε περιπτώσει δικαιώθηκε η διοίκηση, γιατί η οριοθέτηση γίνεται με την εφαρμογή τεχνικών κριτηρίων και με την απαραίτητη τεκμηρίωση. Οπότε, όσα αγαθά κρίνοντα δημόσιο κτήμα, δίνεται, δικαίωμα, δίνεται το δίκαιο στο κράτο. Σε ορισμένε περιπτώσει ε, κρίθηκαν ε, εσφαλμένες οι οριοθετήσει, γιατί δεν ε, ήταν σε δημόσιο κτήμα οι περιοχές αυτές. Ό,τι αφορά τη Φορμεντέρα, το θέμα αυτό κρίθηκε πολλές φορές από το Ανώτατο Δικαστήριο. Και σε όλες τις περιπτώσεις που οριοθετήθηκαν αποφασίστηκε ότι ήταν όντως δημόσιο κτήμα οι περιοχές αυτές, γιατί ήταν είτε σε αμμώδεις περιοχές είτε σε αμμωθήνες. Και μερικές φορές κρίθηκε ότι ήταν αδικαιολόγητη η οριοθέτηση και τότε, σε περίπτωση που το δικαστήριο την έκρινε αδικαιολόγητη, υποχρεώθηκε το Ισπανικό κράτος σε αναθεώρηση αυτής της οριοθέτησης. Πάντως, περισσότερες περιπτώσεις τα δικαστήρια δικαίωσαν τις Ισπανικέ Ισπανικές αρχές. Επαναλαμβάνω, ο νόμος Πυριακτών δεν άρχισε να εφαρμόζεται από το 2008, αλλά από την, εφαρμογή, από την έγκρισή του το 1998. Ούτε εφαρμόζεται αναδρομικά. Υπάρχει ένα μεταβατικό καθεστώς που ισχύει για όσα, όσες ιδιωτικές περνάνε στην κρατική περιουσία και ισχύει το δικαίωμα παραχώρησης. Υπάρχει μια χρονοβόρα διαδικασία που διαρκεί κατά μέσο όρο δύο χρόνια και που δίνει δικαίωμα προσφυγής σε όλους τους θυγόμενους, που δίνει ε, τεκμηριωμένη ενημέρωση στους θυγόμενους, δυνατότητα πραγματογνωμοσύνης επιτόπου με αίτηση του ιδιοκτήτη. Υπάρχουν επίσης δυνατότητες αναθεώρησης αυτής της οριοθέτησης με προσφυγή στα δικαστήρια. Επίσης, δεν θα πρέπει να συγχαίουμε το στόχο αυτού του νόμου περιακτών με την εφαρμογή. Γιατί ο νόμος περιακτών θέλει να αποτρέψει την ε, πολεοδομική συνέπεια αυτής της ε, οικοδόμησης σε μια πολύ στενή ζώνη 100 μέτρων από τις ακτές. Γιατί μέχρι εκεί φτάνει ο νόμος. Άλλωστε πέραν της ζώνης αυτής η αρμοδιότητα για την ε, πολεοδομία ανήκει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Επαναλαμβάνω ότι στόχος του νόμου περιακτών είναι κυρίως η διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Γιατί οι ευάλωτες αυτές παράκτες ζώνες έχουν μια τεράστια αξία, και περιβαλλοντική και πολιτιστική. Μάλιστα όλες οι οικολογικές ε, οργανώσεις στην Ισπανία ζήτησαν την ε, αμετάβλητη εφαρμογή του νόμου περιακτών. Και μάλιστα η σωστή εφαρμογή του νόμου περιακτών επιβεβαιώθηκε όχι μόνο από τα δικαστήρια, αλλά και από άλλους θεσμούς όπως είναι του διαμεσολαβητή, του συνηγόρου του πολίτη. Γιατί έγιναν πολλές αναφορές προς το στο συνήγορο του πολίτη και στις περισσότερες περιπτώσεις κρίθηκε ότι ήταν σωστή η δράση της διοίκησης και κατάλληλη. Εν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι οι Ισπανικές αρχές κατ' εφαρμογή του νόμου ακτών, προσπαθούν να διαφυλάξουν το περιβάλλον των Ισπανικών ακτών και να εξασφαλίσουν την δημόσια χρήση των ε, Ισπανικών παράκτιων ζώνων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο της Ισπανικής Κυβέρνησης. Η τελική συζήτηση για τις αναφορές αυτές αύριο. αφού ακούσαμε και τους αναφερόμενους που θα είναι παρόντες αύριο. Επειδή δεν είχαμε προβλέψει ότι θα μας φάει τόσο χρόνο αυτό το σημείο, σας παρακαλώ να αντιστρέψουμε τη σειρά της ημερήσιας διάταξης. Δηλαδή, οι δύο αιτήσει όπου είναι παρόντες οι αναφερόμενοι από σεβασμό προς τους αναφερόμενους. Να συζητήσουμε πρώτα το σημείο 10. 11 και 12 και μετά θα γυρίσουμε στην ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, ας κάνουμε αυτό. Δύο λεπτά και θα περάσουμε στο σημείο 10.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 Dicevo, riprenderei allora dalle petizioni scritte. Σημείο 10. Αναφορά 313-2007, 670-2009 και 58-2010. Παρόν είναι ο, ο κύριος Νικόλα Στοκ της τρίτης αναφοράς. Είναι παρόν. Έχετε το λόγο κύριε Νικόλα Στοκ. Grazie signor, eh, signor Presidente, signora Presidente. Eh... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτέ, Εδώ εκπροσωπώ την ε, Ένωση Ασοσιασιών Task Force Argentina με εντολή περίπου 180.000 Ιταλοί πολίτες που επένδυσαν σε χρεόγραφα σε ομολογίες τη Αργεντινής το 2001. 4,4 δις δολάρια. μέσα μιας συλλογικής προσφυγής μέσω INGIT που είναι μια οργάνωση της ε, Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον και εκπροσωπούμε και άλλους πολλούς Ιταλούς και Γερμανούς επενδυτές και από άλλα κράτη που έχουν ομολογές χρηστασίου για 5,2 δις δολάρια που φάσαν να μην συμφωνήσουν με την πρόταση ανταλλαγής του 2005 της Αργεντινής και θέλουν να κρατήσουν το χρέος αυτός έναντι της Αργεντινής μέσω εναλλακτικών οδών δικαστικής προστασίας. Ανησυχούμε έντονα με φορέας της ανησυχίας όλων αυτών των Ιταλών πολιτών που υπάρχει κίνδυνος να υποστούν περαιτέρω ζημιά με δράσεις της Αργεντινής κυβέρνησης. Τον περασμένο Οκτώβριο οι Αργεντινοί μερικές εμπορικές τράπεζες Barclays, Citibank και Deutsche Bank με στόχο ορισμένα κερδοσκοπικά επενδυτικά αγγλοσαξονικά κεφάλαια, καμία διαδικασία συμφωνίας δεν έγινε έναντι των ομολογιούχων. Η πρόταση ανταλλαγής του 2005 με όρους που βάσει τον Υπουργό Οικονομίας και θα είναι χειρότερη σε σχέση με την προηγούμενη προσφορά με περιορισμό περίπου στο κατά 65% του αρχικού κεφαλαίου. Προσπάθεια αυτή να αντικατασταθούν οι τίτλοι αυτοί με αξία 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βέβαια, τις λεπτομέρειες ακόμα δεν τις ξέρουμε. Στην αναφορά που έχετε μπροστά σας επισημαίνεται η μη, ε, το μειωμένο κύρος της αργεντινής κυβέρνησης έχει περιθωριοποιηθεί από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κοινότητα και παρότι είναι στους G20 και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Βέβαια, επειδή δεν έχουμε χρόνο, δεν θα τα αναφέρω όλα σε λέει αναφορά, επισημαίνω μόνο ότι η Αργεντινή έχει οικονομικά μέσα. Το δημόσιο χρέος σήμερα είναι κάτω από το 40% του ΑΕΠ. Όταν έκανε το χρεοστάσιο ήταν 120%. Τα αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας είναι πάνω από 48 δις δολάρια. Άρα η χώρα υψηλού κινδύνου συγκρίνεται με τις λεγόμενες high pool indebted country, κακός. Αυτό σημαίνει ότι μία ε, έκδοση ομολογιών της είναι τα έδινεται 7-8 περίπου, ε, ή το διπλάσιο μάλλον από της Βραζιλίας. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει πνεύμα διαφανούς συνεργασίας. Και παραμένει αυτή η κατάσταση χρωστασίου εδώ και 8 χρόνια η προσφορά για την ανταλλαγή για την οποία φαίνεται ότι η Αργεντινή σκοπεύει να καταθέσει τα έγγραφα στο Λουξεμβούργο για πολίτες και κατοίκους άλλων ευρωπαϊκών χωρών με βάση το Prospectus Directive Οδηγία 2003 της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν επενδύσει σε ε, χρεόγραφα της Αργεντινής που δεν διαμένουν σε άλλη χώρα. Με άλλα λόγια δηλαδή, εποφελείται της κοινωτική νομοθεσίας η Αργεντινή και για να μην παρουσιάσει στην Ιταλία ή στη Γερμανία πλήρη περιγραφή και θα περιοριστεί μόνο στη μετάφραση μερικών σελίδων που φυσικά από ό,τι φαίνεται δεν θα περιέχουν όλες τις πληροφορίες για τη νέα προσφορά ανταλλαγή. Οι Ιταλοί επενδυτέ που εκπροσωπούνται και από την Ένωση Μα τη ΕΦΕ και άλλοι Ευρωπαίοι πολίτε, ιδιαίτερα οι Γερμανοί που έχουν χρεόγραφα της Αργεντινής σε χρεοστάσιο θα πρέπει να αποφασίσουν χωρίς να έχουν στα χέρια τους τις αναγκαίες πληροφορίες για να πάρουν μια ε, απόφαση με πλήρη επίγνωση. Καλό την Επιτροπή σας και όλες τις αρμόδιες αρχές, όπως τον ΤΣΕΖ παραδείγματο χάρη, η ανάγκη αυτή της προσφοράς ανταλλαγής να περάσει μέσα από την έγκριση των αρχών εποπτείας των χρηματαγορών της Ιταλίας και της Γερμανίας και τρία επιπλέον σχόλια. Πρώτον, για οποιοδήποτε εκδότη corporate θα μπορεί να μην σέβεται τις αποφάσεις ενός Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να εκπέμπει τις ομολογίες του στο ίδιο κράτος, η ερώτηση είναι ρητορική, αλλά ξέρω στην περίπτωση σε τέριμπους Paribus μπορεί να συμβεί αυτό με την Αργεντινή σε μερικές εβδομάδες. Η Αργεντινή δεν, τήρησε τις, δεν σεβάστηκε τις 450 δικαστικές αποφάσεις γερμανικών δικαστηρίων υπέρ των μικρών ε, ομολογιούχων από την Ευρώπη και άλλες αποφάσεις από το Δικαστήριο της Νέας Υόρκης για Ευρωπαίους πολίτες για να αποκατασταθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνη στην αγορά μεταξύ των αυτών που εκδίδουν τις ομολογίες και αυτών επενδύουν θα πρέπει τα κράτη που ζητάνε την έγκριση και εδώ αναφέρουμε στην Αργεντινή να ε, ε πουλήσουν αυτά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα πέραν των εθνικών συνόρων να γίνει μόνο αν υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τους νόμους και τις αποφάσεις των δικαστηρίων ή των διαιτητικών αρχών έναντι του εκδότη. Δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο η Αργεντινή διαχειρίστηκε το θέμα αυτό της default του χρεοστασίου και σας θυμίζω ότι εκ μέρους του Εκουαντόρ ή το δημοψήφισμα που έγινε στην Ισλανδία να μην πληρωθούν οι Ευρωπαίοι επενδυτές, το ότι δεν υπάρχει αναδιάρθρωση του sovereign default των κρατικών δηλαδή δανείων θα οθήσει και άλλες χώρες για λόγους λαϊκισμού να συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο προς το άμεσο πολιτικό τους πλεονέκτημα βραχυπρόθεσμα αλλά βραχυπρόθεσμα πλήγμα για την ίδια τη χώρα. Αυτό δεν θα έπρεπε να το δέχεται η διεθνή κοινότητα έναντι μιας χώρας που είναι στους G20. Πρέπει να βρεθεί ένα εμβόλιο, κανόνες που να τους αποδέχονται όλες οι χώρες. Και τρίτο, η προστασία της αποταμίευσης των μικρών επενδυτών πρέπει να είναι ο κύριος στόχος του νομοθέτη. Αυτή η προστασία είναι ο στυλοβάτης της σωστής λειτουργίας της οικονομίας. Τα πρόσφατα κρούσματα το αποδεικνύουν αυτό. Πρέπει να υπάρχει εποπτεία του πλούτου, του συνόλου των πολιτών. Αυτό δημιουργεί κοινωνική σταθερότητα. Γι' αυτό τα προβλήματα αυτά χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα πρέπει να λύνονται με διαδικασία αναδιάρθρωσης όπου να εξασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ αυτού που έχει εκδώσει ομολογίες και βρίσκει σε χρωστάσιο και αυτού που έχει επενδύσει. Άλλες λύσεις θα οδηγήσουν σε συγκρούσεις μεταξύ των πολιτών και του κράτους. Σας θυμίζει ένα λατινικό ρητό. Πάκτα sunt servanta. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε κύριε Σοκ. Το λόγο στην Κομισιόν. Στον κύριο Τορνέζε. Στα Ιταλικά. Ευχαριστώ. Θα περιοριστώ στην ε, οδηγία προσπέκτου και πιο συγκεκριμένα στο τι προβλέπεται στα γλωσσικά. Υπάρχει ένα καθεστώς που προστατεύει τους επενδυτές μέσω γλωσσικών διατάξεων που προβλέπει το προσπέκτους να εγκρίνεται στο home member state και μετά να ε, κυκλοφορεί στις άλλες χώρες. Υπάρχει ρητή υποχρέωση η γλώσσα να είναι είτε η γλώσσα της αρμόδιας τοπικής αρχής, host member state, ή η γλώσσα αποδεκτή από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η οδηγία προσπέκτους εγγυάται συνεπώς ότι με βάση μια ανάλυση επιπτώσεων που έγινε πρόσφατα σε σχέση με την αναθεώρηση της οδηγίας αυτής, αποτελεσματική προστασία για τον επενδυτή. Τώρα, για το σημείο που αφορά το summary, τη σύνοψη. Αυτό είναι υποχρέωση να δίνονται επαρκείς πληροφορίες για τους κινδύνους που συνδέονται με την προσφορά αυτή. Και εδώ είναι θέμα εφαρμογής. Η θέση της Κομισιόν στην πρόταση του Σεπτεμβρίου έλαβε υπόψη την ανάγκη αναθεώρησης του περιεχομένου και του τύπου παρουσίασης του summary. Πάντως, οι συνεισφορές και τα στοιχεία που πήραμε από την συνδιαλλαγή μας δείχνουν ότι υπάρχει επαρκής προστασία του επενδυτή. Πρόεδρος, συγγνώμη, αλλά πριν δώσω το λόγο σε συναδέλφους θέλω να κάνω μια διευκρίνηση ως πρόεδρος της Επιτροπής έγραψα μια, ένα σημείωμα στην Κομισιόν, το έστειλα και επισημένω τον προβληματισμό αυτών εδώ των αναφορών και όπως ακούσαμε από τον ε, ανα, λίγο αναφέροντα δεν είναι θέμα γλωσσικό είναι πολύ πιο σοβαρό είναι ένα θέμα χρηματοπιστωτικό, οικονομικό, αφορά εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίους. Και ζώντας τη φάση που ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη με τις χρηματαγορές, η Κομισιόν και ο αρμόδιος επίτροπος θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός με την ουσία και όχι να ασχολείται με τον τύπο των πραγμάτων. Βρίσκω λίγο περίεργη αυτή την απάντηση που δώσατε δεν υπάρχει μια μήνυμου αναφορά, δεν θα έπρεπε, στην επιστολή που έστειλα στην Κομισιόν και να απαντήσετε στα σημεία της επιστολής αυτής. Είναι θέμα χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα, η προσπάθεια μιας προσπάθειας, μια, συγγνώμη, μιας χώρας να καταστρατηγήσει όλους τους διεθνούς κανόνες να χρησιμοποιήσει ύπουλα την νομοθεσία του Λουξεμβούργου στη δική μας ευρωπαϊκή αγορά για να πλήξει εκ νέου Ευρωπαίους πολίτες με μια προσφορά που από ό,τι φαίνεται είναι χειρότερη από την τελευταία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε αναφέρθηκαν σε αυτή τη νέα πρόταση της Αργεντινής και ότι είναι χειρότερη, δηλαδή εξαπατά ακόμα περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και να σηκώσουμε ένα φραγμό και ένα εμπόδιο πριν η αργεντινή κυβέρνηση χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο. Περίμενα κάτι παραπάνω στην απάντηση της Κομισιόν. Κομισιόν. Όντως, είναι ένα πρόβλημα που αφορά τις διεθνείς σχέσεις και αφορά και Και άλλα διεθνή όργανα. Όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, η Αργεντινή δεν βρίσκεται σε πλεονεκτούσα θέση σε σχέση με άλλες χώρες. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ευρωπαϊκά εργαλεία που υπάρχουν και τα οποία προσφέρουν προστασία στον επενδυτή. Υπάρχουν δύο σημεία εδώ πρέπει να προσέξω. Πρώτα είναι το summary που πρέπει να βελτιωθεί στο, στη μορφή την οποία έχει προκειμένου να δίδονται περισσότερες πληροφορίες στον επενδυτή για το default risk, όπως το λέμε, το κίνδυνο χρεοκοπίας ή χρωστησία. Και το δεύτερο, οικονομικό αυτό στοιχείο, η Αργεντινή ας το η διεθνής διάσταση που πρέπει να λάβει υπόψη ο επενδυτής, να λάβει υπόψη ορισμένα προηγούμενα σε σχέση με τη χρήση ενός συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού εργαλείου. Αλλά ως νομοθετικό εργαλείο η προστασία του επενδυτή προστατεύεται. Συγγνώμη, η προστασία του επενδυτή εξασφαλίζεται. με αλλαγή της μορφής και της ουσίας, του περιεχομένου δηλαδή, του summary, έτσι ώστε συνειδητά ο επενδυτής να μπορεί να επενδύσει σε ένα μέσο, χρηματοπιστωτικό μέσο, γνωρίζοντας τους συναφείς κινδύνους. Αυτό αυτή τη στιγμή είναι σε φάση επεξεργασίας στην Κομισιόν. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μποσινάρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας μίλησε για κάποιους μηχανισμούς μέσω των οποίων προστατεύονται οι επενδυτές. Υπάρχει όμως κάτι που είναι πολύ πιο εύκολο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί να μην χρησιμοποιήσει τον διοργανικό διάλογο με την Αργεντινή. Εφόλη τη σύλληση διάλογο με τη χώρα αυτή γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, έθεσε αυτό το θέμα ως προτεραιότητα στις συνομιλίες της με την Αργεντινή. και μέσω του μηχανισμού της αιρεσιμότητας να επιδιώξει μια λύση. Φαίνεται ότι η Αργεντινή δεν έχει αντίστοιχες δεσμευτικές διατάξεις όπως ε, στο κοινοτικό, όπως ισχύουν στο κοινοτικό δίκτυο. Γιατί λοιπόν να μην θέσουμε στις συνομιλίες μας με την Αργεντινή ως προτεραιότητα αυτό το θέμα. Γιατί είμαι βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να προσπίσει καλύτερα τα συμφέροντα των συμπολιτών της αν ε, τους καλύψει γενικά και δεν τους αφήσει τον καθένα στη μοίρα του. Όποιος συνάδελφος θέλει να μιλήσει. Δεν φαίνεται κανείς. Ο Δόκτωρ Σόξ μήπως θέλει να... Έχετε πάλι το λόγο. Είμαι απογοητευμένος ειλικρινά κυρία Πρόεδρε από τον παρέμβαση της, του εκπροσώπου της Κομισιόν. Ε, πάλι καλά για αυτό που δεν αγόρασε ομολογίες της Αργεντινής. Διαφορετικά δεν θα ήταν τόσο τυπικό στην απάντησή του. Η Αργεντινή έκανε ό,τι ήθελε. Καμία παρέμβαση δεν υπήρξε εκ μέρους των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων ή της Κομισιόν να προασπίσει τις εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτών που επένδυσαν σε κρατικές ομολογίες της Αργεντινής, όχι σε ιδιωτικέ επιχειρήσεις μικρές. Και όταν μιλάμε για εγγύηση των επενδύσεων των bonds στην Αργεντινή, η εγγύηση ήταν τι ήτανε. Η Αργεντινή πρόσφερε το 35% της ονομαστικής αξίας. 35% εγγύηση, αν και γράφεται παντού, και έχω δει τα προσπέκτους που λέει ότι για 50 χρόνια η Αργεντινή δεν χρεοκόπησε όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Μάλλον χρεοκόπησε. Σας καλώ λοιπόν, όχι εγώ, η πρόεδρος πρέπει να το κάνει, να ξαναδούμε το θέμα στην ουσία του. 180.000 Ιταλοί, πάνω από 100.000 άλλοι, εκ των οποίων 70.000 Ισπανία έχασαν ένα σωρό λεφτά. Πήγαν σε δικαστήρια. Προσφυγή κατά της Αργεντινής και η Αργεντινή δεν πλήρησε ούτε καν τα δικαστικά έξοδα. Εγγυήσεις που ότι η Αργεντινή ότι τηρεί τους κανόνες των, του χρηματοπιστωτικού συστήματος αυτό δεν αληθεύει. Πρόεδρος. Εγώ δεν εξέφρασα την μη ικανοποίησή μου ακόμη. Πάντως έχω γράψει επιστολή στον Επίτροπο Μπαρνιέ όπου ζητάω απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα και απάντηση δεν πήρα. Το θέμα παραμένει ανοιχτό για να πάρουμε, μέχρι να πάρουμε μια απάντηση στις ερωτήσεις που θέσαμε και που τη συμφωνήσαμε με τις επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων. Και όπως είπε ο Σνέφος Μποσινάρο, καλούμε την Κομισιόν στη συνάντηση του Μαΐου μεταξύ της Κομισιόν και της Αργεντινής Κυβέρνησης Στη συνάντηση αυτή και μέχρι τότε η Κομισιόν θα πρέπει να δεσμευτεί να δει πιο ζεστά αυτό το θέμα που αφορά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και βάζει σε σκληρή δοκιμασία το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα που ήδη έχει πληγεί σοβαρά από τις, τα πρόσφατα γεγονότα. Αν οι συνάδελφοι συμφωνούν, προτείνω αυτό ως λύση. Παραμένει στην ημίρησα διάταξη η αναφορά αυτή. Και περνάμε στο επόμενο σημείο, το 11. 1143 του 2008 του Ερικ Σανίτας και Φρανσουάντε Τρουαγέ. Ο πρώτος αναφέρον έχει το λόγο, Ερικ Σανίτας. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για το ότι δέχτηκε την αναφορά μας και μας έδωσε τη δυνατότητα να σας αναλύσουμε την περίπτωση. Όταν υποβάλαμε την αναφορά μας, επιμείναμε ε, στο πρόβλημα που δημιουργεί η κατάσταση των, ε, των εκδόσεων κρατικών ομολόγων. Και ενδιαφερθήκαμε κυρίως για τα δομημένα προϊόντα. Φαίνεται ότι δικαιωθήκαμε γιατί οι δυσκολίε που αντιμετώπισαν χώρε όπω η Ελλάδα που ακολούθησε την Ισλανδική κρίση φερικιότητες και μάλλον προηγείται της κρίσης πολλών ακόμη και κοινοτικών χωρών, επιβεβαιώνουν τις πιο απεσιόδοξες προσεγγίσεις ε, και αμφισβητούν την τυφλή βεβαιότητα της ασφάλειας των ε, δημόσιων χρεογράφων. Θα πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί ο τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης ε, των κρατών που εκδίδουν τέτοια ομόλογα. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ήταν αρκετά πρωτοπόρο και ψήφισε ένα κείμενο μαζί με την αναφορά αυτή, ζητώντα ε, πλαισίωση των δραστηριοτήτων των rating agencies, μετά μάλιστα την εξέλιξη και της αμερικανικής νομολογίας που αμφισβήτησε την ατιμορρησία αυτών των ε, οργανισμών. Θα πρέπει να, έχουμε, να, να ασκηθεί ένας αποτελεσματικός έλεγχος στις στους οργανισμούς αυτούς αξιολόγησης και να τροποποιηθούν ε, οι κανονισμοί λειτουργίας αυτών των ε, οργανισμών. Το κεντρικό σημείο για μας της νέας αυτής ρύθμισης αφορά την ε, υποχρέωση των οργανισμών να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους και που σχετίζονται με την εφαρμογή των μεθόδων τους. Και στην παλιά και στη νέα νομοθεσία οι ίδιοι οι οργανισμοί σε με μέλημα την ανεξαρτησία των οργανισμών να κρίνουν ποια είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να λάβουν υπόψη και που έχουν στην ε, διάθεσή τους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής έναντι της απροθυμίας μιας, ενός οργανισμού να λάβει υπόψη στοιχεία που, τις κοινοποιούνται, του Φαίνεται από την υπόθεση ότι υπάρχουν σημαντικές δυσλειτουργίες στη λειτουργία αυτών των οργανισμών. Την περίπτωση του Moody's, που αναφέρει στη μεθοδολογία ότι η, δυνατό, η, βούληση της πληρωμής είναι το κλειδί της ανάλυσης των κρατικών ομολόγων. Βέβαια, η περίπτωση της άνησης της Ρωσίας να πληρώσει δείχνει ότι δεν είναι δεδομένη μια τέτοια ισχυρή βούληση για πληρωμή. Και μάλιστα η ανάλυση του προβλήματος από τη Standard Poor's είναι χαρακτηριστική. Ο οργανισμός αυτός θεωρεί ότι Υπάρχουν κάποια αποπευθέντα χρέη που έχουν εκδοθεί από προηγούμενη κυβέρνηση και που δεν λαμβάνονται υπόψη στο παθητικό της, ε, της τωρινής κυβέρνησης. Τότε ε, αποσύρουμε το καθεστώς του χρεοστασίου αν ε, το ζήτημα δεν διευθετηθεί σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Αν λοιπόν το ζήτημα δεν έχει ε, λυθεί σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, αγνοείται το απαράγραφο του δημόσιου χρέους. Οπότε, σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται εδώ η αρχή της συνέχεια των κρατών και το γεγονός ότι ε, απορρίπτεται αυτό το χρέος θεωρείται φυσιολογικό. Θεωρείται φυσιολογικό λοιπόν να αποφασίσει η κυβέρνηση αν θα ε, αποπληρώσει ένα χρέος που έχει συνάψει η προηγούμενη κυβέρνηση. Η Standards Poor's λοιπόν ε, στο μηχανισμό που χρησιμοποιεί δεν θεωρεί τον, το χρεοστάσιο ως την έλλειψη της, της πληρωμής ενός ε, τόκου, ενός κεφαλαίου. Ενώ η Moody's θεωρεί ότι θεωρεί χρεοστάσιο οποιαδήποτε πληρωμή δεν έγινε ή είναι υπερήμερη σε ό,τι αφορά τον τόκο ή το κεφάλαιο. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία αυτών των ε, οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα κρατικά ομόλογα οι rating agencies ε, θα πρέπει να συμβάλλουν στην ασφάλεια δικαίου και στην εφαρμογή του δικαίου. Με τη συμπεριφορά τους όμως αυτή φαίνεται ότι θα ενισχύσουν τον κρατούντα σκεπτικισμό. Αποφασίσαμε λοιπόν ε, να ζητήσουμε τις ε, αναγνωρισμένες μεθόδους αναγνώρισης. Στραφήκαμε λοιπόν στο γραφείο ΕΣΕΟ, e στο γραφείο ΑΝΤΕΟ που είναι μέλος του ΣΑΗ και εκπροσωπείται από τον κύριο Πιέρα Μπέρ, που θεωρεί ότι ε, ένα τέτοιο χρέος δεν μπορεί να, να αποτιμηθεί σε λιγότερο από 8.000 ε, ευρώ. Και μάλιστα με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή μπορεί να φτάσει και στα 40.000 ευρώ. Δεν γνωρίζουμε όμως ε, το εύρος αυτού του Θέλουμε λοιπόν ε, να λάβουμε οποιαδήποτε μέτρα που να ε, πιστοποιούν την ύπαρξη αυτού του χρέους, κάτι που μας αρνούνται οι rating agencies. Οι οργανισμοί αυτοί στηρίζονται σε κάποια στοιχεία που έδωσε η Ρωσική Ομοσπονδία και που είναι φαλκιδευμένα και μάλιστα αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη γιατί αυτά τα κρατικά ομόλογα εκδόθηκαν από μια κυβέρνηση που καμουφλάρισε τους λογαριασμούς της. Μάλιστα, τα κρατικά ομόλογα στηρίχθηκαν σε πλαστά έγγραφα. Κάτι που δεν μας διαβεβαιώνει ότι στο μέλλον η Ρωσία θα είναι διαφανής σε τέτοιες εκδόσεις κρατικών ομολόγων. Δεν θα πρέπει τα κρατικά ομόλογα να βρίσκονται στο απειρόβλητο μηχανισμών ελέγχου. Θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη αυτών των κρατικών ομολόγων. Από το 2001, μία ένωση κομιστών τέτοιων χρεογράφων της Ρωσίας άσκησαν προσφυγή στην γαλλική δικαιοσύνη ε, επικαλούμενοι ότι δεν ελήφθη υπόψη από τη Ρωσία το προηγούμενο χρέος τότε η προσφυγή αυτή θεωρήθηκε σχεδόν βλάσφημη. Αυτό έκρινε η γαλλική δικαιοσύνη, απορρίπτοντας την προσφυγή, θεωρώντας ότι ε, είναι ε, αβάσιμη η αγωγή, παρόλο που ο στόχος ήταν εύλογος. Ε, γιατί θεωρήθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν κάποιες διαδικασίες εις βάρος τρίτων που μπορεί να οδηγήσουν σε ζημία τους. Αυτή μάλιστα η συστηματική προσπάθεια προάσπισης των συμφερόντων των πιστοληπτικών οργανισμών από τις πλευράς των δικαστηρίων είναι πραγματικά αξιολύπητη. Δεν θα πρέπει η δράση αυτή να χρησιμοποιηθεί απλώς για να είναι καλές οι σχέσεις με τη Ρωσία. Γιατί δυστυχώς έτσι έχασε μια μεγάλη ευκαιρία ε, αξιοπιστίας η γαλλική δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ. Grazie, do la parola al secondo petente. Δεύτερος αναφέρον Φρασάντε Τουραγίου. Σας παρακαλώ να είστε λίγο πιο σύντομος αν γίνεται. Εκπροσωπώ την Ένωση Σκρίπτα Ρούσια Μάνα του Βελγίου εκπροσωπεί τους κατόχους ε, κρατικών ρωσικών ομολόγων. Σε λίγε εβδομάδε, κύριε και κύριοι, η Ρωσία θα εκδώσει κρατικά ομόλογα αξίας 17,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα χρήματα θα τα δανειστεί από αποταμιευτέ που θα έχουν εμπιστοσύνη στην ομοθεσία και στην ε, ειλικρίνεια των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ε, ε, ικανότητας χωρίς να ξέρουν ότι θα δανείζονται τα, θα δανείζουν τα χρήματά τους σε ένα κράτος που ουσιαστικά φαλκιδεύει τα στοιχεία του, του λογαριασμούς του και προσπείται μια υγιή δημοσιονομική διαχείριση που δεν έχει. Μάλιστα, οι κάτοχοι τέτοιων ομολόγων που εκδόθηκα πριν από το 1917 γνωρίζουν ότι η φαλκίδευση τέτοιων στοιχείων είναι μια πραγματικότητα που σήμερα η Ευρώπη προσποιείται ότι ανακαλύπτει με την περίπτωση της Ελλάδας. Χάρη στην ευρηματικότητα των χρηματοπιστωτικών, χρηματο, ε, χρηματοπιστωτικών φορέων η Ελλάδα κατάφερε να αποκλείσει από τα λογιστικά της στοιχεία ένα σημαντικό αποθετικό, δίνοντας ε, απατηλή εικόνα για την οικονομική της κατάσταση και τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων της. Και μάλιστα αυτή η απατηλή κατάσταση διευκολύνθηκε από τη συγκαταβατικότητα των rating agencies. Μάλιστα η κρίση των ε, subprimes ε, έδειξε πόσο εσφαλμένες ήταν οι αξιολογήσεις τέτοιων τοξικών παραγόγων. Και μάλιστα το παράδειγμα της Ελλάδας δείχνει ότι αυτό που έκαναν οι οργανισμοί για ορισμένα ε, διαρθρωμένα προϊόντα μπορούν να γίνουν και για δημόσιο χρέος. Ποιος θα προειδοποιήσει όμως τους αποταμιευτές και τους ε, επενδυτές. Πολλά αναφέρθηκαν για την αναφορά μας. Για παράδειγμα, μας είπαν το χρέος για το οποίο ζητάτε αναγνώριση έχει παραγραφεί. Τα ομόλογά σα είναι αντίκε που εκδόθηκαν από ένα αυτοκρατορικό κράτος που έχει περάσει στη λύθη. Γιατί λοιπόν αυτοί, οι οργανισμοί δολίω ε, παρακάπτουν τον κανόνα της διαδοχής των κρατών, όπως έκανε η Standard και Poor's που στις 23 Φεβρουαρίου έγραψε ότι πάυση πληρωμής ε, του χρέους μιας προηγούμενης κυβέρνησης που είχε ε, εκδώσει το χρέος πριν από πολλά χρόνια και μάλιστα μετά από μια αποπομπή του, της επόμενης κυβέρνησης δεν είναι ενδεικτικό της αφαιρεγγιότητας ε, των τωρινών χρεών και μάλιστα τα ομόλογα της κυβέρνησης Παπανδρέου θα είναι έγκυρα μόνο αν η επόμενη κυβέρνηση τα πληρώσει. Πραγματικά διαφωνούμε με τα κριτήρια της Standard και Poor's στις 16 Νοεμβρίου 2009 και όχι 1909 αλλά 2009 κυρίες και κύριοι ε, σε ένα γαλλικό δικαστήριο η Ρωσική Ομοσπονδία επικαλέστηκε και μάλιστα με επιτυχία τον κανόνα της διαδοχής των κρατών για να απαιτήσει την απόδοση της του Ορθόδοξου Καθεδρικού Ναού της Νίκαιας με το επιχείρημα ότι αρχικά είχε αγοραστεί με τον προϋπολογισμό του αυτοκρατορικού ε, κράτους. Γιατί λοιπόν η γαλλική δικαιοσύνη δέχεται την εφαρμογή αυτού του κανόνα της διαδοχής για την περίπτωση της ε, επιστροφής του καθεδρικού ε, ναού της Νίκαιας, αλλά όχι για την ε, αποπληρωμή των παλιών κρατικών ομολόγων. Μας είπαν επίσης ότι η επίσημη αναγνώριση της παύσης πληρωμής ε, ουσιαστικά εξυπηρετεί τα συντεχνιακά συμφέροντα κατόχων παλιών τσαρικών ε, χρεογράφων. Φυσικά και θέλουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα, γιατί οι οργανισμοί ε, αξιολόγηση πιστοληπτική ικανότητα δεν κάνουν τη δουλειά του και τα κράτη εθελοτυφλούν. Μάλιστα δεν είμαστε οι μόνοι που θυγόμαστε. σα είπα πριν από λίγο ότι η Ρωσία θα εκδώσει νέα κρατικά ομόλογα. Θα αφήσουμε λοιπόν τους Ευρωπαίους αποταμιευτές να αγοράσουν στο, ε, στην, στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου τέτοια χρεόγραφα ενός κράτους ε, που ενώ έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές συγκαλύπτει και καμουφλάρει τους λογαριασμούς και δεν τις πληρώνει. Πώς έγινε η αξιολόγηση του ισολογισμού της Ρωσίας και δεν βρέθηκαν ίχνη από, τα, από τις αξιώσεις που δεν έχουν πληρωθεί. Το ίδιο δεν συνέβη και με την Γαλλία, με την Ελλάδα, συγγνώμη που φαίνεται ότι παραπίσε τους λογαριασμούς της. Δεν ήξεραν λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία οι οργανισμοί ε, αξιολόγησης. Δεν είναι μόνο η Ρωσία και η Ελλάδα που καμουφλάρει τα στοιχεία και τους λογαριασμούς. Ας μην ξεχνούμε και την Κίνα που οι απλήρωτες αφιλές της έχουν ε, εγγραφεί στο χρηματιστήριο του Παρισιού. Μην μας λέτε λοιπόν ότι κατέχουμε αντίκες δεν ε, έχουν παραγραφεί όλα αυτά τα χρέη, τότε γιατί η γαλλική κυβέρνηση ετοιμάζεται την άνοιξη να διαπραγματευτεί με την κινέζικη κυβέρνηση ένα ανύπαρκτο υποτίθεται χρέο. Λυπούμε λοιπόν από όλε τι χώρε ε, να ανοίξουν τα κοιτάπια τους και να ελεγχθούν από τις ευρωπαϊκές αρχές. Ζητούμε έλεγχο των χρηματοπιστωτικών φορέων για να αποφύγει οποιοδήποτε ε, κίνδυνος προσποίησης ή παραποίησης. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποια βέβαια ρευστά ληξιπρόθεσμα χρέη που η ύπαρξή τους έχει βεβαιωθεί από αποταμιευτές καλόπιστους ε, εφόσον έχει αναλυθεί ανάλυση και η βούληση πληρωμής των εκδοτών. Το προηγούμενο Ιανουάριο, ο κύριο Σαλμούνια ζήτησε από την Ευρωστάτ να αποκτήσει και ελεκτικέ αρμοδιότητε που το 2005 δεν κατάφερε να πάρει για να μπορέσει να επαληθεύσει τα στοιχεία που υποβάλλονται από τι χώρε μέλη. Στι 15 Φεβρουαρίου, ο κύριο Γιόνκερ ε, ζήτησε συγγνώμη από όλο τον κόσμο γιατί άφησε στη Eurogroup, στην οποία προείδρευε, να αρνηθεί στη Eurostat την επέκταση των αρμοδιοτήτων το 2005. Ο κύριος Φερχόφστατ είπε θα ήθελε να μάθει πώς ολόκληρη η πολιτική αλυσίδα και η διοικητική αλυσίδα από την Αθήνα στις Βρυξέλλες, περνώντας από τη Φραγκφούρτη, κατάφερε να αγνοήσει όλο αυτό το καμουφλάρισμα των ελληνικών δημοσίων λογαριασμών. Θέλουμε λοιπόν όλα αυτά τα διαβήματα, αλλά να μην περιοριστούμε μόνο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να περιλαμβάνουμε όλα τα κράτη που εκδίδουν ομόλογα που μπορούν να αγοράσουν οι Ευρωπαίοι αποταμιευτέ. Δεν θα πρέπει να διακινδυνεύεται έτσι η Ευρωπαϊκή Αποταμίευση. Μην ξεχνάτε και την Ισλανδία. Και μην ξεχνάτε τι έγινε με τους Ολλανδούς και Γάλλους αποταμιευτές που δάνεισε στην Ισλανδία. Δεν μπορούμε να κάνουμε πλάτες ε, στο καμουφλάρισμα των δημοσίων λογαριασμών. Θα πρέπει να δώσουμε μάχη για εκατομμύρια ε, αποταμιευτές που θέλουν να αγοράζουν χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί καλόπιστα. Επίσης ε, θα πρέπει το μη αναγνωρίσιμο δημόσιο χρέος να περιλαμβάνεται στα παθητικά στοιχεία ενός κράτους και αυτό θα πρέπει να αναλυθεί ε, για να μην, να καταστραγηθούν τα δικαιώματα όλων αυτών των αποταμιευτών. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται η χορήγηση συγκαταβατικής βαθμολογίας από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ιδιαίτερα για βέβαια χρέη, ρευστά και ληξιπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως ανέφεραν οι αναφέροντες, η ε, τα γραφεία αξιολόγησης του πιστοτικού κινδύνου δεν ε, ελέγχονταν μέχρι τώρα και πράγματι βρίσκονται στην καρδιά της παρούσας ε, οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 2009 το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν το νέο πλαίσιο για να ρυθμίσουν ε, τα, τα γραφεία αυτά, διότι μέχρι τώρα δεν ρυθμίζονταν. Με το νέο αυτό λοιπόν πλαίσιο, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εισήγαγαν ε, υποχρεωτική καταχώρηση των γραφείων αυτών ε, και υπόκεινται σε αυστηρές προϋποθέσεις ώστε να αποφευθούν οι κίνδυνοι σύγκρουσης ε, ενδιαφερόντων. διασφαλίζεται οι υπηρεσίες αξιολόγησης του πιστοτικού κινδύνου να λειτουργούν με διαφανή τρόπο. Οι κανόνες αυτοί θα εφαρμοστούν πλήρως από το Δεκέμβριο του 2010. Δεν ισχύουν ακόμα. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να τηρούνται διότι τα γραφεία αξιολόγηση του πιστοτικού κινδύνου θα ε, εποπτεύονται από Ευρωπαίους και εθνικούς επόπτες. Θα ε, εγκαθιδευτεί λοιπόν ε, σύντομα ε, ε, ένα νέο καθεστώς, το οποίο θα αντιμετωπίσει πολλά από τα θέματα που αναφέρετε εσείς στην αναφορά σας. Επίσης, ε, στον κανονισμό υπάρχει διάταξη που ζητάει από την Κομισιόν να αξιολογήσει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012, σε δύο χρόνια δηλαδή, θέματα όπως είναι η ε, υπερβολική ε, εξάρτηση από τις ε, αξιολογίες πιστοτικού κινδύνου που ισχύει σε κάποιες από τις χώρες μας και επίσης όσον αφορά το μοντέλο το οποίο δημιουργείται από τα γραφεία αξιολόγηση του πιστοτικού κινδύνου. Σε δύο χρόνια λοιπόν ε, θα πρέπει να γίνει η αξιολόγηση από την ε, θέση σε ισχύ του κανονισμού αυτού. Θα αξιολογηθεί λοιπόν εάν υπάρχουν ακόμα προβλήματα στην ε, σχετική αγορά. Ο στόχος του νομοθέτη με τον, την πρόταση αυτή ήταν να λύσει τα περισσότερα από τα προβλήματα. Όσον αφορά το παρελθόν, τα γραφεία αυτά δεν ρυθμίζονταν. Υπήρχε κώδικας δεοντολογίας οι αρχέ όμω δεν είχαν τη δυνατότητα να τις επιθεωρήσουν και να επιβάλλουν κυρώσεις. Με τον νέο κανονισμό θα έχουν οι αρχέ τη δυνατότητα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος να έφερε τέτοιο λόγο. Η κυρία Γκρουνή. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν απάντησε στους αναφέροντες, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε, να μείνει η αναφορά ανοιχτή, να μην κλείσει. Να δούμε τι έγινε το Δεκέμβριο του 2010, να μείνει ανοιχτό για το 2011 και το 2012. Και θα θέλω να ακούσω οι αναφέροντες ικανοποιήθηκαν με την απάντηση της Κομισιόν. Πάντως θεωρώ ότι η αναφορά πρέπει να παραμείνει στο τραπέζι. Χρειαζόμαστε ακόμα δύο χρόνια για τον να αρχίσουν αποτελεσματικά οι έλεγχοι. Μποσινάρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με την ε, συνάδελφο συντονίστρια του ΕΛΚ να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή μετά από δύο χρόνια να ξαναδούμε ποια θα είναι η καταγγελότερη λύση, κυρίως για να αποφευθούν παρόμοιες κρίσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Θα παραμείνει η αναφορά στο τραπέζι προκειμένου να αρχίσουν να εφαρμόζονται αυτά που μας ανάφερε η Κομισιόν. Οι αναφέροντες θέλουν να προσθέσουν κάτι. Ναι. Χωρίς να υπερβάλλω, ερχόμαστε από μια κατάσταση πλήρους αναρχίας που κάνω ό,τι θέλανε οι αξιολογικοί αυτοί, οι οργανισμοί αξιολόγησης. Αυτό που κατάλαβα από το μέχρι στιγμή είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, γιατί διαβάζοντας το κείμενο του Κοινοβουλίου, δεν ξέρουμε τι θα βγει από το κείμενο αυτό. Οι προθεσμίες τέλος 2010, αρχές 2011 είναι πω προθεσμία. Είναι σωστό να παραμείνει στο τραπέζι αναφορά. Να δούμε τι θα δώσει το νέο σύστημα. Θέλω μετά από ένα ή δύο χρόνια να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω εξ ονόματο του συναδέλφου. Αυτά, αυτή είναι η δική μου γνώμη, πρόεδρο. ξανά με του αναφέροντες και περνάμε στο επόμενο σημείο. Η αναφορά 12. 11-20 του 2009. Μάρκο Γκριφίνι, εξόμενος οργάνωσης Αμίτσι bambini Ο Μάρκο Γκριφίνι αν είναι παρόν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής σας. Το Αμίτσι bambini είναι μια ε, διεθνής οργάνωση προς προστασία του δικαιώματος των παιδιών σε θέματα υιοθεσία. Τι θέλουμε με την αναφορά αυτή. Ζητάμε να, ξανανοίξει, να ξανανοίξουν οι διεθνείς ε, από τη Ρωμανία, όπως εξάλλου το ζήτησε μια, ένα κείμενο της ε, συνθήκης του Ηνωμένων Εθνών για τα μου του παιδιού, όπως στην παράγραφο 55 αναφέρεται, η Επιτροπή ζητάει, το συγκεκριμένο κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους νόμους και τις εγγύησει των νομικών για την διεθνή υιοθεσία σύμφωνα και με την συνθήκη της Χάγης για την προστασία των ανηλίκων να αποσύρει το μορατόριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή που είναι εμπόδιο στην πλήρη εφαρμογή του άρθρου 21 της Συνθήκης για τα Δικαιώματα των Ανηλίκων του 89 των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, για ποιο λόγο κάναμε αυτή την αναφορά. Εμείς ως ε, κίνημα των γυναικών που, ε, συγγνώμη, γονέων που δράσει σε 30 χώρε τις διεθνείς υιοθεσίε το θεωρούμε ω την τελευταία λύση. Τελευταία λύση για τα παιδιά αυτά που τα έχουν πετάξει δύο φορές. Τα έχει πετάξει η αρχική οικογένειά τους και τα έχει πετάξει και η οικογένεια η πρώτη που τα υιοθέτησε. Η χώρα μάλλον. Έτσι ώστε να δράσει επικουρικά η νομοθεσία, όπως λέει η συνθήκη της Άγιας να προβλέψουμε την εγκατάλειψη, να βοηθήσουμε δηλαδή την οικογένεια να μην εγκαταλείψει το παιδί και μετά να προωθήσουμε τις διεθνείς υιοθεσίες. όπου θα παίρνουν μέρο όλε οι οργανώσει. Η μόνη χώρα στην οποία δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια αντίστοιχη ένωση είναι η Ρουμανία. Δρούμε εκεί από το 1987, κάναμε ένα ρωμανικό ίδρυμα, πρωτενε Δουλέψαμε δηλαδή προκειμένου να υπάρξουν οι όροι τα παιδιά αυτά να καταλήξουν σε μια οικογένεια. Γι' αυτό μα παραξένεψε πολύ το ότι η χώρα αυτή που την αγαπάμε έκλεισε τι διεθνεί υιοθεσίε, έκλεισε αυτή τη δυνατότητα για χιλιάδε παιδιά να έχουν μια οικογένεια. Τα νούμερα τα ξέρουμε. Τι παθαίνουν τα παιδιά αυτά που βγαίνουν από τα διάφορα ιδρύματα όταν κλείνουν το 18ο έτος ηλικίας. Το 30% περίπου αυτοκτονούν, περνάνε στην πορνεία, στην εγκληματικότητα. Πολλά σκάνδαλα. Βέβαια υπήρξαν και πολλά σκάνδαλα που τα καταγγείλαμε και στις ρωμανικές αρχές και αποκοινούμε τις ρωμανικές αρχές. Αλλά όπως κάναμε και με μεγάλες άλλες οργανώσεις σε πολλές άλλες χώρες, εμείς θέλουμε να υπάρξουν οι όροι νομιμότητας, μέγιστες οροφές και η Ρωμανία την είχε τη δυνατότητα αυτή να αλλάξει την νομοθεσία και να μπει στην νομιμότητα. Διεθνώ, ακολουθώντας το παράδειγμα μια άλλη χώρα κοντινής τη τη Βουλγαρίας, που ήταν τα ίδια χρόνια στι ίδιες συνθήκε. αλλά επέλεξε εντελώ διαφορετικό δρόμο η Βουλγαρία σήμερα. Είναι μια χώρα που έχει ένα πολύ ωραίο νόμο, ένα πολύ καλό παράδειγμα στην Ένωση πώ μπορεί να διαχειριστεί κανεί απολύτω νομίμω το θέμα τη διεθνούς υιοθεσίας. Δυστυχώ η Ρουμανία και λυπάμαι που το λέω αυτό σε Ευρωπαίου πολίτε, είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει απαγορεύσει τις διεθνείς υιοθεσίες. Είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν αναγνωρίζει την διεθνή υιοθεσία ως δικαίωμα του εγκαταλειμμένου ανήλικου. Ωστόσο έχει επικυρώσει τη συνθήκη της Άγιας που ορίζει ρητά ότι η διεθνής υιοθεσία μπορεί να δώσει τη δυνατότητα μια μόνιμη οικογένεια σε ανήλικους παιδιά που δεν έχουν βρει μια κατάλληλη οικογένεια στη χώρα προέλευσης. Έχουμε στοιχεία πολύ πολύ πρόσφατα από το ιστοσελίδα της Λόρα που είναι το επίσημος φορέας στη Ρουμανία. Μιλάει για το Σεπτέμβριο του 2009 τα νούμερα. Σήμερα έχουν, υπάρχουν περίπου 70.000 παιδιά. 24.000 είναι σε ιδρύματα και 45.000 περίπου είναι σε άλλου είδους μονάδες. Εξ αυτών οι 12.682 παιδιά κρίθηκαν υιοθετήσιμα. Οι ρωμανικές οικογένειες που τη 2008 ήταν 2.815. Από τις 2.815 ρωμανικές οικογένειες που πήραν πιστοποίηση να υιοθετήσουν ένα παιδί, υιοθέτησαν μόνο, υιοθέτησαν μόνο οι 885 οικογένειες και το 80% πήρε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. Τα, οι, επόμενοι, οι, οι υπόλοιποι 11.000 ανήλικοι υιοθετήσιμοι με βάση τις ρωμανικές αρχές, τι θα γίνει με αυτούς. Η πρότασή μας είναι σιγά σιγά να ανοίξει η διεθνής υιοθεσία. Γερασπέτσια τι είναι, είναι τα ανήλικα παιδιά με ειδικά χαρακτηριστικά που συνήθως δεν επιλέγονται από μια οικογένεια της. Είναι παιδιά πάνω από, 7 παιδιά, από ηλικία 7 ετών, είναι παιδιά που έχουν αδέλφια, είναι παιδιά με αναπηρίες. Ζητάμε βαθμία να ανοίξει αυτό με διμερείς συμφωνίες που θα υπογραφούν με τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τους περισσότερους Ρωμάνους μέσα στη χώρα κατοίκους να οριστούν οι κανόνες με τις διμερείς συμφωνίες. Τελευταίο παράδειγμα ήταν με τη Ρωσική Ομοσπονδία, έτσι ώστε η διεθνής υιοθεσία να γίνεται με διαφάνεια και σωστά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Εκπρόσωπος της Κομισιόν, η κυρία Ντελούκα. Ευχαριστώ. Όπως, περι... Όπως την περιέγραψε την κατάσταση, ο αναφέρον. Έτσι είναι και είναι γνωστή στην Κομισιόν. Το 2009 κάναμε μία μελέτη για τη διαδικασία υιοθεσία στην Ευρώπη και στις 27 χώρες και δημοσιεύτηκε η μελέτη αυτή παράλληλα με τη μελέτη του Ευρωκοινοβουλίου. Έχουμε δύο πρόσφατες μελέτες λοιπόν για την υιοθεσία στην Ευρώπη. Τι μας λένε αυτές οι μελέτες, ότι η Ρουμανία είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που de facto κατάργησε τη διεθνή υιοθεσία. Με ένα νόμο του 2004 πάρξε να ισχύει τον Ιανουάριο του 2005. Υπάρχει μια μικρή δυνατότητα ε, τέτοιων υιοθεσιών, αλλά περιορίζεται μόνο σε παππούς ή γιαγιάδες βιολογικούς ενώ του παιδιού που, ζει στο, που ζουν στο εξωτερικό αυτοί μπορούν να υιοθετήσουν τα εγγόνια τους και οι συγγενείς μέχρι τρίτο βαθμό, δηλαδή οι και θείες. Ε, αυτό δεν είναι πραγματική υιοθεσία. Πέντε χρόνια ζωής αυτού του νόμου και αρχίζουμε να βλέπουμε και δειλές κινήσεις στη Ρουμανία. Η ώρα που είναι ο αρμόδιος φορέας στη Ρουμανία, το ανάφερε ο αναφέρον. Τον Οκτώβριο μετά από πολλές συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και με την UNICEF που παρακολουθεί το θέμα έκανε πρόταση αλλαγής του νόμου. Να ξαναρχίσουν οι διεθνείς υιοθεσίες παιδιών άνω των 7 ετών, άνω των 6 ετών, συγγνώμη, παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας ή που έχουν κάποια συγκεκριμένη εθνική καταγωγή, πιο συγκεκριμένη Ρώμα, παιδιά, που δύσκολα υιοθετούνται στη Ρουμανία. Αυτή η πρόταση έγινε στον Πρωθυπουργό απορρίφθηκε αμέσω. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. «30 Νοεμβρίου του 2009 η Κομισιόν και με το Συμβούλιο της Ευρώπης μαζί οργανώσαμε μια διεθνή διάσκεψη στο Στρασβούργο όπου συζητήθηκε το θέμα και της εθνικής υιοθεσίας και δηλαδή η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που αναθεώρησε την προηγούμενη του 1974 και τη δεύτερη μέρα, 1η Δεκεμβρίου, συζήτηκαν τα θέματα της διεθνούς υιοθεσία με βάση τη συνθήκη της Χάγης, ιδιωτικού δικαίου, που είναι ένα διεθνές κείμενο, συνέχεια του, της Συμφωνίας του 83 με βάση όλη, του οποίου όλες οι ευρωπαϊκές χώρες με εξαίρεση την Ιρλανδία που ακόμα δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση αυτή, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες την έχουν προσυπογράψει και η Ρουμανία. Ο στόχος αυτής της ε, σύμβασης είναι να εφαρμοστεί το άρθρο 21 των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του, παιδιού. Τι λέει το 21? Ότι η οθεσία είναι ένας τρόπος να βρεθεί οικογένεια για παιδιά που δεν έχουν, αλλά θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην, εθνικό, ε, στην εθνική οικογένεια που υιοθετεί, αλλά αν προς το συμφέρον του παιδιού ε, λύση είναι η ε, διεθνής υιοθεσία και αυτό ισχύει. Η Κομισιόν παρακολουθεί το θέμα αυτό της διεθνούς υιοθεσίας θα πάρει μέρος στην Ειδική Επιτροπή, Συνδρίαση ειδική Επιτροπής στη Χάγη τον Ιούνιο. Το πρόβλημα της Ρουμανίας είναι πολιτικό, δεν είναι νομικό. Η Ρωμανία έκανε μια πολιτική επιλογή. Κατάργησε τις διεθνείς υιοθεσίες. Και όπως είπε ο εκπρόσωπος της UNICEF, στη διάσκεψη που σας ανάφερε του Στρασβούργου. Αυτή η επιλογή θα μπορούσε να είναι σωστή, αλλά το 2005 για να δείξει η χώρα ότι θέλει να βάλει πέρας στην έλλειψη διαφάνειας, στο ότι υπήρχαν κρούσματα διαφθορά στην υιοθεσία κλπ. Ένα θετικό μήνυμα της Ρουμανίας. Και η Βουλγαρία έκανε το ίδιο πράγμα. Ε, εισήγε ένα μορατόριο στην διεθνή ε, υιοθεσία. Αλλά στο μεταξύ η Βουλγαρία έχει ψηφίσει ένα νέο νόμο, ο οποίος λειτουργεί και οι διεθνείς υιοθεσίε ε, γίνονται πια με τήρηση των διεθνών αρχών και κυρίως προς το συμφέρον του παιδιού. Αυτό δεν γίνεται στη Ρουμανία. Τι να κάνει η Κομισιόν. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε μια πολιτική επιλογή μιας χώρας μέλος. Ο αναφέρον αναφέρθηκε σε διμερείς συμφωνίες. Είναι δυνατές τέτοιου είδους συμφωνίες. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κοινοτική νομοθεσία, γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, άρα τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν μεταξύ τους διμερείς συμφωνίες. Ευπρόσδεκτο αυτό. Αλλά οι διμερείς συμφωνίες απαιτούν δύο. Άρα πρέπει να συμφωνεί και η Ρουμανία. Μέχρι στιγμής, από ό,τι ξέρουμε, αυτό δεν συμβαίνει. Παρακολουθούμε λοιπόν εκ του σύνεγγυς της εξελίξης και σε ελπίσουμε ότι πολιτικά θα αλλάξει η κατάσταση. Εμείς εντό εισαγωγικών υποδείξαμε στην απάντησή μας, στην αναφορά, ότι ενδεχομένως ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου θα βοηθούσε. Το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει βέβαια. Γι' αυτό ευχαριστώ. Πρόεδρος. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την απάντηση αυτή της Κομισιόν. Μακάρι να σας ακολουθήσει το Κοινοβούλιο Μποσινάρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μπονασέρα κύριε Γκριφίνη, Πρόεδρε της Ένωσης Φίλοι των Παιδιών. Συνεχίζω στα ρωμανικά. Θα ήθελα να να εκφράσω την περιφρόνησή μου προς το τελευταίο σχόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί σχεδόν αγγίζει τα όρια της προσβολής προς τη Ρουμανία. Θα ήθελα να μείνουμε στη νομική βάση και στα νομικά επιχειρήματα σε ό,τι αφορά την προστασία των παιδιών στη Ρουμανία. Γιατί η Ρουμανία έχει γίνει ε, ευρωπαϊκή υπόθεση σε ό,τι αφορά την υιοθεσία. Το 1992 η Ρουμανία εξήγαγε και μάλιστα εδώ παραθέτω έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάνω από 3.000 παιδιά το χρόνο. Δηλαδή πάνω από το 1,9% του συνόλου των παιδιών που γεννιόνταν στη Ρουμανία. Μεταξύ 1997 και 2001 με βάση τα στατιστικά στοιχεία. Και δεν μιλώ για τα αγνοούμενα παιδιά, για τα παιδιά που εξαφανίστηκαν, που δεν περιλαμβάνονται καν στα Μητρώα δηλαδή. Μεταξύ 1997 και 2001 η Ρουμανία ενέκρινε πάνω από 9.300 ε, διεθνείς υιοθεσίες, κάτι που αποτελεί τραγωδία και όνειδος για τη ρουμανική ιστορία. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ επίσημα τις Βρυξέλλες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ε, συνέβαλαν στο να εξαλειφθεί αυτή η μάστιγα στη Ρουμανία. Γι' αυτό και από το 1997 συστηματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμεινε στο πρόβλημα των διεθνών υιοθεσιών και των περιπτώσεων διαφθοράς και δωροδοκίας που διαπιστώθηκαν σε, τέτοιου, σε τέτοιους περιπτώσεις διεθνούς νομοθεσίας. Αυτό ήταν αγκάθι στις σχέσεις Ρουμανίας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε το θέμα σε υπουργικό επίπεδο και σε μία μόνο νύχτα πάνω από 400 ντοσιέ χάθηκαν στο Ρουμανικό Υπουργείο γιατί ζητήθηκε επίσημα έρευνα της Europol και της Interpol. Υπήρχε τέτοιος βαθμός δωροδοκίας και διαφθοράς που φαίνεται ότι κάποιος πλήρωσε για να εξαφανιστούν εντός εισαγωγικών όλοι αυτοί οι φάκελοι με τις ε, περιπτώσεις των παιδιών. Και φτάσαμε και στη, στα δικαστήρια, αλλά πολλές φορές στα δικαστήρια επέλεγαν ποια παιδιά θα στέλνονται στις διεθνείς ομοθεσίες. Και είπε επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση, stop, φτάνει πια, θα πρέπει να αναλυθεί κάποια δράση. Και αυτό φάνηκε το 1999, όπου ζητήθηκε επανειλημμένως από τη ρουμανική κυβέρνηση να να δώσει προτεραιότητα στην προστασία του παιδιού. Δεν ήταν η Ρουμανία που αποφάσισε κάτι τέτοιο. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Ρουμανική κυβέρνηση να επιβάλλει την προστασία των παιδιών. Και λυπούμε που περνάω απότομα από τα ρουμανικά στα αγγλικά. Λοιπόν, αυτή η θέση, αυτό το επιχείρημα περιλήφθηκε σε όλες τις εκθέσεις πρόοδου και σε όλες τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι που μπήκε η, Ευρωπαϊ... η Ρουμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα η πιο σημαντική διακήρυξη ήταν ε, το ανακοινωθέν τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό και θα ήθελα να υπενθυμίσω την εκπρόσωπο, στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην ξεχνά τις προηγούμενες δηλώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα ανακοινωθέντα τύπου. Αναφέρθηκε λοιπόν στην έκθεση προόδου για τη Ρουμανία που, του 2005 ότι η νέα ε, ρουμανική νομοθεσία για τα δικαιώματα του παιδιού και την υιοθεσία που τέθηκε και σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2004 είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη συνθήκη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συμπληρώνει τη μεταρρύθμιση στο θέμα της προστασίας του παιδιού. Παρόμοια πρακτική ε, εφαρμόζεται και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη και η διακρατική υιοθεσία δεν, ε, θεωρείται ως μέτρο προστασίας του παιδιού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγο τροποποίηση αυτή της ε, νομοθεσία στη Ρουμανία. Αυτά λέει η έκθεση προόδου και παρακολούθηση της Ρουμανίας τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρεται λοιπόν εδώ ότι η Ρουμανία δεν ε, σέβεται και παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία. Και για να αποφευθούν οποιασδήποτε παρεκτροπές από το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, να σας πω κάτι που είπε ο Γκίντερ Φερχόγεν τότε, που ήταν αρμόδιος επίτροπος για τη διεύρυνση και μετά έγινε και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είπε έναν εξάρτητο πάνελ από εμπειρογνώμονες οικογενειακού δικαίου, συγκροτήθηκε και πάλι στα ρουμανικά ο κ. Μποστινάρου. Και τι είπε τελικά αυτό το έγγραφο, που διαβάσατε όλοι και που βρίσκεται στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορείτε να το διαβάσετε. Αναφέρεται λοιπόν σε αυτό το έγγραφο ότι η ρουμανική νομοθεσία σέβεται πλήρως τις ευρωπαϊκές διατάξεις, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Επίσης αναφέρεται ότι η Διεθνής νομοθεσία, η διακρατική νομοθεσία θα πρέπει να αποτελέσει εξαιρετικό μέτρο, ε, να συνοδεύεται από περιορισμούς και πραγματικά να είναι ίστατο μέτρο, μέτρο εκτάκτου ανάγκης ή ασχάτου ανάγκης. Και αυτές ε, ε, οι ρυθμίσεις εγκρίθηκαν χάρη στο Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γουίντερμπορ που είναι φιλελεύθερη, όχι σοσιαλίστρια, αλλά όλα αυτά τα έκανε για την Ρουμανία και για τα παιδιά της Ρουμανίας. Τώρα δηλαδή θα καταστρέψουμε όλες τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλες τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παρήχε και τεχνική βοήθεια και χρηματοοικονομική βοήθεια στη Ρουμανία και πολλές συμβουλές και τώρα να λέμε ότι θα πρέπει να γίνονται πια ακόμη, για μια ακόμη φορά ελεύθερα οι διεθνείς υιοθεσίες και πάλι στα ρουμανικά. Κύριε Ματζόνη, στην Ρουμανία στις 4 Φεβρουαρίου του 2004 είχαμε ένα σκάνδαλο που απασχόλησε και πολύ καιρό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο δήμαρχος του Βουκουρεστίου, σοσιαλιστής, ε, εξέδωσε ένα ολόκληρο κατάλογο με δεσμεύσεις, γιατί ασκήθηκε τεράστια πίεση και μάλιστα η τότε κυβέρνηση είχε δεχθεί κατ' εξαίρεση ε, στο πάγωμα των διεθνών ε, υιοθεσιών κάποιες υιοθεσίες και τότε υπόθηκε κάτι που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Τζον Κέρι, ο Λιονέζο Πέ, ο Χωσέ Μαρία Σνάρο, τότε Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Ρουμάνο Πρόντι, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Μπερλουσκόνη, ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας το καλοκαίρι του 2003 είχε στείλει επιστολή στον Ρουμάνο Πρωθυπουργό Αναστάση ζητώντας ε, κατεπηγόντω να επιτρέψει ε, την ε, παρεκτροπή από το μορατόριου και για να αποφευθεί αυτή η τραγωδία και να προστατευτούν οι ευρωπαϊκές αξίες. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν υπέβαλε τροπολογίες ε, στη Ρουμανική νομοθεσία για, την, ε, για τον περιορισμό των διεθνών υιοθεσιών. Σε καμία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε καμία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν τροποποιήθηκε αυτή η πρόταση. Σήμερα μόνο ακούμε κάτι τέτοιο. Και πρώτη φορά ακούμε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα θα ήθελα να αρχιοθετήσουμε την αναφορά αυτή, γιατί είναι αδικαιολόγητη. Η Επιτροπή μας θα πρέ... έχει αρχιοθετήσει και άλλες αναφορές για τις υιοθεσίες στη Ρουμανία. Υπάρχει δηλαδή προηγούμενο. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε το λόγο σε κάποιον που αυτή την επονίδιστη περίοδο της ρουμανικής ιστορίας όπου είχαμε εξαφάνιση παιδιών, παιδιών που χρησιμοποιήθηκαν για εμπόριο οργάνων. Υπήρξαν πολλές μορφές κατά της Ρουμανίας. Παιδιά που έγιναν βορρά του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος ή διαφόρων εγκληματικών κυκλωμάτων. Να δώσουμε το λόγο και στην εκπρόσωπο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προστασίας των ε, παιδιών που πρόσφατα δημοσίευσε το βιβλίο «Ρουμανία μόνο για εξαγωγή». Δυστυχώς είναι τραγική και άβολη αλήθεια που αναφέρει, όπως είπε η Γκαλγκόρ, δυσάρεστη αλήθεια, αλλά μιλά για την πραγματικότητα που ίσχυσε αυτή τη τραγική δεκαετία στη Ρουμανία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μποστινάρου. Μποστινάρου. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μανσόνη. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να διαβάσω τον κατάλογο που δημοσίευσε σήμερα η ε, ρουμανική κυβέρνηση. Το Ρουμανικό Γραφείο για τις υιοθεσίε εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τις πιέσεις ε, που έχουν ασκήσει κάποιες ε, διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις στα ευρωπαϊκά φόρουμ για να αναγκάσει τη Ρουμανία να ξανανοίξει τις ε, διεθνείς ε, υιοθεσίες. Σήμερα δημοσιεύτηκε αυτό. Κατά τη διάρκεια του 2009 και μέχρι τώρα, το Γραφείο Υιοθεσιών της Ρουμανίας ε, προσπαθεί να εντοπίσει λύσεις για να κινητοποιήσει τις διεθνείς υιοθεσίες, δεδομένου του ότι εδώ και κάποια χρόνια ο, ο αριθμός οικογένειών που θέλουν να υιοθετήσουν παιδί είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό παιδιών προς Δεν έχουμε δηλαδή παιδιά για υιοθεσία. Όλα τα βήματα που έχει αναλάβει το Γραφείο Υιοθεσιών της Ρουμανίας επικεντρώνονταν στη διευκόλυνση της διαδικασίας της ε, ε, υιοθεσίας ε, προς του παιδιού. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού οικογενειών που ήθελαν παιδιά υιοθεσία, προτεραιότητα της, ε, του, του οργανισμού μας είναι να προωθήσει ε, καλές πρακτικές για υιοθεσία, ε, η οποία να είναι προς όφελος των παιδιών και να σέβονται τις αρχές που αναφέρονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού με στόχο να ε, λαμβάνεται υπόψη ε, κατά την εκπαίδευση του παιδιού η ε, εθνοτική, θρησκευτική και πολιτιστική του ταυτότητα. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε σημαντικές αμφιβολίες σχετικά με την αναφορά που τέθηκε στην Μέση διάταξη σήμερα, διότι το θέμα που συζητάμε θα έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και καιρό. Κυρία Μανσόνη, θα ήθελα προσωπικά να σας ρωτήσω γιατί μπήκε η αναφορά αυτή στην ημερήσια διάταξη σήμερα, καθότι έχουμε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2005, το 2006, το 2008 σε παρόμοιες ε, ε, αναφορές ε, που έλεγε ότι η Ρουμανία σέβεται το διεθνή νόμο περιοθεσία. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπέβαλα προσφυγή στον, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Η συζήτηση της αναφοράς αυτή σήμερα μου, για μένα είναι σαφώς χάρη προς ε, την ε, πρόεδρο της ε, Επιτροπής, διότι ο, τον, ο αναφέρον έχει την ίδια εθνικότητα με την πρόεδρο. Ελπίζω να κλείσει λοιπόν αυτό και θα ήθελα να σας πω ότι είμαι κατά ενός ψηφίσματος για το θέμα αυτό. τα, τα ρουμανικά μέλη της ε, Επιτροπής ΠΕΤΗ προέρχονται από διαφορετικές ε, πολιτικές ομάδες. Δυστυχώς όμως όλοι συμφωνούμε μεταξύ μας όσον αφορά τα παιδιά της χώρας μας να σας θυμίσω τι συνέβη με τα ρουμανικά παιδιά που δόθηκαν προς εθεσία στο εξωτερικό ανάμεσα στο 1997 και το 2004. 10.936 παιδιά υιοθετήθηκαν από ξένες ε, οικογένειες από τα, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ισπανία, την ε, Ιταλία, τη Δανία και την ε, Ελβετία. Ε, περίπου 1.300 ε, παιδιά δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε πια, δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Η Βαρόνη ε, Έμα Νίκολσον, η συγγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Ρουμανία επικρίνει τη Ρουμανία για εμπορία παιδιών. Η Ρουμανία λοιπόν αποφάσισε να θέσει μορατόριο για να σταματήσει τις διεθνείς υιοθεσίες, ε, κάτι για το, προς το οποίο την κάλεσε ε, διεθνείς οργανισμοί και τον Ιανουάριο του 2005 ε, τέθηκε σε ισχύ νόμος για τις διεθνείς υιοθεσίες και δημιουργήθηκε το, Γραφείο, το Γραφείο Διεθνών Υιοθεσιών της ε, Ρουμανίας. Στις εκθέσεις για τη Ρουμανία και την ε, Βουλγαρία αναφέρεται το θέμα των δικαιωμάτων του παιδιού και αναφέρεται ότι οι υιοθεσίες γίνονται ε, σε συμφωνία με, την, ε, με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Επίσης, σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ, η Ρουμανία προσυπάρουσε την σύμβαση αυτή καθώς και τη Σύμβαση τη Χάγης του 1993. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Υιοθεσία Παιδιών αναθεωρήθηκε ε, στο Στρασβούργο το, 2008. Σύμφωνα λοιπόν με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών στη, για τη διαδικασία της υιοθεσία, ε, το συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να είναι η πιο σημαντική πτυχή, το οποίο σημαίνει ότι κανένα άλλο συμφέρον οικονομικό, πολιτικό, ε, ή του ατόμου που υιοθετεί δεν θα πρέπει να να, αποτελεί προτεραιότητα σε σχέση με το συμφέρον του παιδιού. Ε, θέλουμε να αποτρέψουμε του ανθρώπου που θέλουν να υιοθετήσουν παιδιά από τη Ρουμανία επειδή αυτό, κάτι τέτοιο είναι πιο εύκολο. Δεν είναι πιο εύκολο. Η διεθνή υιοθεσία δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση για το παιδί. Ε, η νομοθεσία της Ρουμανίας ε, τροποποιήθηκε το 2004. Το παιδί μπορεί να υιοθετηθεί από ε, ε, συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού, ε, τους ε, παππούδες του ή θείους και θείες. Θέλουμε τώρα να διευρύνουμε το, την κατηγορία των παιδιών που μπορούν να υιοθετήσουν το παιδί για να συμπεριλάβουμε για τους συγγενείς τέταρτου βαθμού, καθώς και Ρουμάνους συγγενείς στο εξωτερικό. Εάν οι προθέσεις σας ήταν τόσο καλές, θα γνωρίζατε ότι στη Ρουμανία ο αριθμός αιτήσεων ξεπερνάει τον ε, αριθμό των παιδιών που προς υιοθεσία. Ο αριθμός ε, των οικογενειών που θέλουν να υιοθετήσουν είναι σχεδόν διπλάσιος ε, του αριθμού των παιδιών, που είναι, των παιδιών προς υιοθεσία. Είμαι κατά μιας, ενός ψηφίσματος για το θέμα αυτό, εφόσον η, η ρουμανική νομοθεσία συμφωνεί με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μιλάμε για ε, ψήφισμα. Μέχρι στιγμή όλα τα μέτρα που ελήφθησαν από ε, τι Ρουμανικέ Αρχέ υποστηρίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Μπιλ Πόξ, ε, ο Πρωθυπουργό της Ρουμανίας, είπε πέρσι ότι οι διεθνεί Ρουμανίας, συγγνώμη, ότι οι διεθνεί υιοθεσίε δεν θα ξανανοίξουν και έτσι θα παραμείνει η κατάσταση προ το παρόν. Τέλο, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γκριφίνη γιατί ξαφνικά δείχνει τέτοια ανησυχία για τα ρουμανικά παιδιά. Οι Ρουμανικέ αρχέ και τα δικαστήρια για θέματα υιοθεσία δεν μπορούν να παρακολουθούν στενά όλα τα παιδιά που έχουν υιοθετηθεί στο εξωτερικό. Η μη κυβερνητική οργάνωσή σας ε, με τον ε, ε, περιορισμένο προπολογισμό μπορεί πράγματι να παρακολουθεί όλα τα ρουμανικά παιδιά στο εξωτερικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφα Θα απαντήσω αμέσως αντιλαμβάνουμε την προσωπική ενδιαφέρον ε, τη συναδέλφου Μπασέσκου. Δεν με φύγει προσωπικά. Εγώ ε, νομίζω ότι κάνω ασκώ το έργο μου και αυτό μπορεί να το κρίνουν και οι συνάδελφοι για όλους τους τελευταίους αυτούς μήνες. Η ανάφορα αυτή γιατί έμεινε στη μεσαία να έχουμε κλείσει με άλλε παρόμοιε αναφορέ. Διότι αυτή εδώ η αναφορά από την Ένωση που εκπροσωπεί ο κύριος Γκριφίνη μας έφερε ανησυχητικά στοιχεία σε γνώση. Αυτό κρίναμε ότι με, με εκατοντάδες ορφανά Περίπου το 80% των πορνών που έρχονται στην Ιταλία είναι κάτω των 18 ετών και είναι από τη Ρουμανία. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία. Η διαμαρτυρία του Ηνωμένων Εθνών, επιστολή του Ιουνίου, Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καλεί με τις συστάσεις προς τη Ρουμανία ζητάει παρέμβαση της Ρουμανίας σε σχέση με τον νόμο αυτό που συζητάμε, γιατί θεωρεί ότι είναι αντίθετο με τον συμφέρον των ε, ανηλίκων στη Ρουμανία και παραβιάζει τα δικαιώματα του παιδιού και του εφήβου, όπως ορίζονται στην ε, συνθήκη για τα δικαιώματα των ανηλίκων που έχει υπογράψει η Ρουμανία. Αυτό είναι ένα τμήμα των λόγων για τους οποίους οδήγησαν την Προεδρία και τους συντονιστές να ξαναβάλουμε στην εμερήσια διάταξη αυτή την αναφορά. Δεν έχουμε την παραμικρή πρόθεση να παρεύουμε στα εσωτερικά της κυβέρνησης της Ρουμανίας. Θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι μπροστά σε τέτοιες καταγγελίες και τέτοια νούμερα. Και όπως είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν έχουμε πολιτική και ηθική φυσικά υποχρέωση να παρέμβουμε με ένα ρόλο διαιτητικό προσφέροντας τις καλές μας υπηρεσίες. Η συνάδελφος Στόγια. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την αναφορά αυτή. Σε πρώτο πλάνο βάζω τα παιδιά όλα τα παιδιά της Ευρώπης, άρα και τα παιδιά της Ρουμανίας που είναι παιδιά της Ευρώπης, πέρα από τους ελάχιστα αποδεκτούς υπενιγμούς της συναδέλφου Μπασέσκου και τον τόνο με τον οποίο απευθύνθηκε στην ε, Επιτροπή μας. Αγαπητή Δεσποινής Μπασέσκου, όλα αυτά είναι πολύ εύκολα να αντιστραφούν ως ισχυρισμοί γιατί υπάρχει θέμα συμφερόντων εδώ. Κανένας μας εδώ μέσα δεν πρέπει να κατηγορεί τον άλλον να μιλάει για κακές προθέσεις. Οι μη κυβερνικέ οργανώσει που ασχολούνται με τις διεθνείς υιοθεσίε είναι αξιέπαινες. Το έργο τους το ασκούν με, μεγάλη, μεγάλες θυσίες και με πολλή αγάπη για τα παιδιά προς το συμφέρον του παιδιού και συχνά μεταξύ μιας χώρας και τη άλλη χώρα δημιουργούνται δεσμοί αλληλεγγύη με τις υιοθεσίε αυτές. Δεν έχω μόνο κατά νου τη Ρουμανία. Εμείς οι Ιταλοί είχαμε υιοθετήσει παιδιά και από άλλε χώρες. Δημιουργούνται δεσμοί στοργή, ανταλλαγή, αμοιβαία γνώση. Γι' αυτό βρίσκα, βρήκα προσβλητικού τους ισχυρισμούς τη συναδέλφου. Και το λέω προς, τώρα προς τον συνάδελφο Μποσινάρο. Όταν η Ρουμανία υποστηρίχθηκε από την Ένωση, το Ευρωκοινοβούλιο, την Κομισιόν και είχε το θάρρος να παγώσει προσωρινά την κατάσταση, να κάνει ένα μορατόριο. Όντω, γιατί η κατάσταση ήταν τραγική και πολύ σωστά κηρύξατε μορατόριο. Και όλοι το δεχτήκαμε. Γιατί όταν μιλάμε για εθεσία, το πρώτο είναι το παιδί να εξασφαλίσει μια οικογένεια, μια βοήθεια πέραν εκμετάλλευσης ή οποιοδήποτε κινδύνου. Οι διεθνείς εθεσίες λοιπόν πρέπει να γίνουν με συνθήκες ασφάλειας για το μέλλον του παιδιού που να βρει μια οικογένεια που θα το υποδεχτεί και να υπάρχει η παραμικρή υποψία εκμετάλλευσης. Αυτό το μαρατόριο λοιπόν ήταν χρήσιμο. Και όλοι το δεχτήκαμε. Όμως Ήταν μεν τραγική η κατάσταση τότε. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν χρόνια. Περιμένω γιατί θέλω ο συνάδελφος ε, ο να με ακούσει. Αυξήθηκε ο ρυθμός των ορφανών. Μιλάμε για ορφανά χωρίς οικογένεια όχι αυτά που είχαν μια οικογένεια που, ήταν, που τα έβαλε στο ορφανοτροφείο και αυτό οδήγησε σε εκμετάλλευση κλπ. Παιδιά που δεν έχουν πια οικογένεια. Και ξέρω ότι υπάρχουν αιτήματα υιοθεσία, αλλά όπω και στην Ιταλία, οι γονεί που θέλουν να υιοθετήσουν θέλουν ένα παιδί πολύ μικρό, για να το εκπαιδεύσουν οι ίδιοι, υγιέ, ενώ υπάρχουν παιδιά που δεν είναι πολύ μικρά πια που χρειάζονται ειδική θεραπεία ή περίθαλψη, γιατί έχουν δυσκολίε. Άρα η οικογένεια που θέλει να υιοθετήσει ένα τέτοιο παιδί έχει πολύ ισχυρά κίνητρα προσωπικά δικά τη. Ξέρω ότι στην Ιταλία υπάρχουν γονεί που δεν έχουν την καταλληλότητα να υιοθετήσουν και ταυτόχρονα θέλουν ένα παιδί. Πάρα πολύ μικρό, αν είναι δυνατόν και πολύ όμορφο και πολύ υγιέ, δεν είναι αυτό το πνεύμα αυτού που υιοθετεί. Α δούμε τα παιδιά που δεν τα ζητάνε εντό εισαγωγικών γιατί χρειάζονται ειδική φροντίδα και περίθαλψη. Αν λοιπόν η κατάσταση σε πολλές χώρες απαιτεί ως τελευταία λύση την διεθνή υιοθεσία, γιατί για μια προσπάθεια με την αρχική οικογένεια, μετά μέσα στη χώρα, με την πολιτική να μείνουν τα παιδιά στη χώρα τους. Αν όμως υπάρχει παρόλα αυτά η ανάγκη και υπάρχει διάθεση από το εξωτερικό, γιατί να αποκλείσετε την διεθνή υιοθεσία με όλες τις εγγυήσεις που χρειάζονται, όχι όπου να είναι και σε όποιον να είναι, γονιό. Αν υπάρχουν χώρες που θέλουν να κάνουν κάτι διμερός, να το μελετήσουμε. Ήρεμα το θέμα, οι δύο κυβερνήσεις, οι αντίστοιχες ενώσεις, οργανώσεις, τι θέλω να πω, ας βρούμε έναν τρόπο να δώσουμε απάντηση. Κανένας δεν κατηγορεί, κανένας δεν αμήνεται εδώ μέσα. Δεν μιλάμε για μη κυβερνητικέ οργανώσεις που εμπορεύονται παιδιά. Μιλάμε για μη κυβερνητικέ οργανώσεις ελέγξιμες, ελεγμένες, που συνεργάζονται. Στην Ιταλία έχουμε πολλούς Ρουμάνους που ζουν στην Ιταλία. Θα μπορούσε λοιπόν να ήταν μια χώρα με την οποία θα μπορούσε να υπάρχει μια προτιμησιακή σχέση. Και οι Υπουργοί Εξωτερικών Κυβερνήσεων της Αριστεράς, που είναι το κόμμα το το ζήτησαν, δεν είναι ένα κόμμα που το ζήτησε. Είναι ένα αίτημα όλων όσοι στην Ιταλία είναι υπέρ της μετανάστευσης και της ρωμανικής μετανάστευση που δεν την επικρίνουν. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να αποκατασταθεί έστω μια διμερής επαφή, γιατί να μείνουν τα παιδιά για πάρα πολλά χρόνια στα ορφανοτροφία, για καμία χώρα, ακόμα και για την πιο πλούσια, δεν είναι η καταλληλότερη λύση, γιατί μετά ενηλικιώνονται και δεν έχουν καμία δυνατότητα ένταξη στην κοινωνία. Δέστε την καλή βούληση, την καλή προαίρεση που υπάρχει πίσω από την πρόταση αυτή. Προτείνετε κάτι θετικό, όχι με τον τόνο όλο κατηγορίες των συναδέρφων. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι θα κάνουμε. Όχι. Συζητάμε και η πλειοψηφία που ψηφίζει. Ζητά από τους συναδέρφους που είναι λιγότερο αυθαρχικοί στις διατυπώσεις τους να το σκεφτούν το θέμα με αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος Μαρτίνες. Εγώ κυρία Πρόεδρε, επουδενή δεν εστερνίζομαι τις επικρίσεις που ασκήθηκαν ε, εις βάρος σας. Τα πράγματα εμφανίζονται στην σε διάταξη στην ώρα τους, ως με το ρυθμό και με τη σειρά που υποβάλλονται. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι υπήρξε κακή προαίρεση από οποιονδήποτε. Θα ήθελα να μιλήσω καταρχήν με διπλή ιδιότητα. Καταρχήν ως παλέμαχος ευρωβουλευτής, αλλά και ως παλέμαχος φίλος της Ρουμανίας. Και νομίζω ότι οι βετεράνοι παλέμαχοι έχουμε υποχρέωση να καταθέτουμε τη μαρτυρία μας. Και καλό είναι να ακουστεί κάποιο ε, μη Ρουμάνος. Να σας υπενθυμίσω ποια ήταν η κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από 5-6-7 χρόνια. Τότε έγινε μια τεράστια διεθνής κινητοποίηση και μια εκστρατεία που έφερνε τη Ρουμανία σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι η εκστρατεία εκείνη ήταν υπερβολική και ξεκινώντα από κάποια πραγματικά αξιοθρύνητα στοιχεία έδινε μια χείριστη εικόνα για τη Ρουμανία, παρουσίαζε τη Ρουμανία σαν κόλαση. Μέχρι και ορισμένε φωτογραφίε ήταν α, παραποιημένες. Δημιουργήθηκε όμως μια τόσο τεράστια κινητοποίηση που ακόμη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εξέταζε την υποψηφιότητα της Ρουμανίας για ένταξη χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα, στους φίλους της Ρουμανίας και στους υπόλοιπους. Και οι φίλοι της Ρουμανίας προσπαθήσαμε να πιέσουμε τους Ρουμάνους φίλους για να δεχτούν μία ε, προϋπόθεση, τουλάχιστον ένα μορατόριουμ για να κλείσει το πρόβλημα. Και να κλείσει και το στόμα κάποιων που πραγματικά δημιουργούσαν ένα κολοσιαίο σκάνδαλο και προπαγάνδα εις βάρος της Ρουμανίας, που σε καμία περίπτωση δεν ήταν δικαιολογημένη σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις, γιατί ε, μερικές φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε αμερικανικά συγκεκριμένα περιοδικά ήταν πλαστές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστάτησαν ε, σε αυτή την ε, κατάσταση και εμείς παροτρύναμε και σχεδόν ε, επιβάλαμε στη Ρουμανία αυτό το μορατόριο. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να σεβαστούμε τη Ρουμανία, να σεβαστούμε τη ρουμανική κυβέρνηση και να αφήσουμε τη ρουμανική κυβέρνηση να αποφασίσει ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανασταλεί αυτό το μορατόριο. Δεν είναι δική μας δουλειά. Γιατί κάτι που είπαμε πριν από λίγα χρόνια και μάλιστα με στεντόρια φωνή και σχεδόν κάνοντας εκβιασμό στη Ρουμανία. Ας μην ε, κάνουμε τον εκβιασμό προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν μπορώ εγώ τώρα να ζητήσω από τις Ρουμανικές αρχές να διακόψουν ή να αναστείλουν το μορατόριο. Εγώ θεωρώ ότι οι Ρουμανικές αρχές είναι υπεύθυνες και περισσότερο από τον καθένα μας έχουν μέλημά τους το καλό των παιδιών, περισσότερο ακόμη και από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Νομίζω ότι αν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή που ενδιαφέρεται περισσότερο για το καλό των ρουμανικών παιδιών, είναι η ρουμανική κυβέρνηση. Ποιο άλλο ενδιαφέρεται περισσότερο για τα παιδιά τη Ισπανία από την Ισπανική κυβέρνηση. Οπότε και η Ρουμανική κυβέρνηση το ίδιο ενδιαφέρεται για το αγαθό των, και τα συμφέροντα των παιδιών τη Ρουμανία. Δεν είμαι πατερναλιστή εγώ. Δεν μπορώ να, να δίνω μαθήματα σε ορισμένες χώρες, ενώ δεν δίνουμε μαθήματα σε άλλες χώρες. Γιατί υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν θα τολμούσαμε να τους κάνουμε μάθημα και κήρυγμα και να τους πούμε αλλάξε την νομοθεσία σας. Εγώ είμαι από εκείνου που πιστεύω ότι δεν υπάρχουν παλιά και νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι είμαστε ίσοι και αξίζουμε σεβασμό και αξιοπρέπεια. Ας περιμένουμε λοιπόν από τις, αρμονικ... από τις αρχές που είναι οι αρμόδιες να λάβουν υπόψη αυτά που ακούσαμε, τα επιχειρήματα των ΜΕΝ και των ΔΕ, αυτά που ισχυρίζονται τα Ηνωμένα Έθνη και με όλα αυτά τα στοιχεία θα αποφασίσουν ποια είναι η κατάλληλη στιγμή, πότε είναι σκόπιμο, θα αποφασίσουν οι ρουμανικές αρχές, πότε είναι σκόπιμο και σωστό για τα παιδιά που το συμφέρον τους λαμβάνουν υπόψη να αναστείλουν το μορατόριο και προσοχή. Σε τέτοιου είδου ζητήματα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί σίγουρα υπάρχουν μη κυβερνητικέ οργανώσει με μεγάλη γενεοδορία, αλλά πριν από λίγου μόνο μήνε είχαμε μία μη κυβερνητική οργάνωση που όλοι θα βάζαμε το χέρι μας στη φωτιά για αυτήν, που είδα, είδαμε ότι στην ΑΕΤ είχαν απαγάγει 60 παιδιά, υποτίθεται για το καλό τους. Από τα παιδιά όμως αυτά που για το καλό τους ε, απήχθηκαν. Μας είπαν τώρα για τη Ρουμανία ότι από αυτά τα παιδιά έβγαζαν όργανα για μεταμόσχευση. Αυτό αναφέρθηκε για τη Ρουμανία τότε, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδόν επέβαλαν στη Ρουμανία το μορατόριο ή την κατάργηση της δυνατότητας της διεθνούς υιοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε και πολύ προσεκτικοί και να σεβαστούμε τη χώρα αυτή. Και να δείξουμε εμπιστοσύνη ότι μια χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην οποία λειτουργεί και ισχύει το κράτος δικαίου, είναι υπεύθυνη να κρίνει πότε είναι σκόπιμο και πότε δεν είναι σκόπιμο να αναστείλει το συγκεκριμένο μορατόριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βαλιάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από όλα όσα ακούσαμε εδώ πέρα, θα ήθελα να πάμε εγώ πίσω στην αρχική συζήτηση. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα λόγω μιας αναφοράς Ιταλικής μη κυβερνητικής οργάνωσης για να μιλήσουμε για τις διεθνείς υιοθεσίες στη Ρουμανία. Το νόμο για τις διεθνείς υιοθεσίες. Δεν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε την προστασία του παιδιού στη Ρουμανία. Ναι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε αυτό οι Ρουμάνοι λέμε ότι έχουμε έναν από τους καλύτερους νόμους στην Ευρώπη, ένα παράδειγμα ε, προς μίμηση. Δεν βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τα ορφανά της Ρουμανίας, δεν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε καν για τις πόρνες στην Ιταλία. Δεν βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την οδηγία ελεύθερης κινητικότητας των Ευρωπαίων πολιτών και τον τρόπο που η Ιταλία επιλέγει να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή αυτή οδηγία. Βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε τον νόμο περί διεθνούς υιοθεσία στην Ρουμανία. Η Ρουμανία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφάσισε, έλαβε μόνο της απόφαση για το θέμα αυτό. Εάν η Ρουμανία αποφασίσει να κλείσει τις διμερείς διαπραγματεύσεις με, ε, τα άλλα, με κράτη, αυτό είναι θέμα της Ρουμανίας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν με εκπλήσει ότι έχουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη σήμερα ε, και το έθεσε στην ημερήσια διάταξη η πρόεδρος της Επιτροπής. Δεν διαφωνώ με αυτό, ε, αλλά με εκπλήσει πάρα πολύ η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα. Διότι παραδέχεται ότι δεν υπάρχει νομική βάση για την προσφυγή αυτή. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο εκπρόσωπός της, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνο, επιλέγει λοιπόν να κάνει πολιτικές δηλώσεις, διότι πρόκειται για πολιτική δήλωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο εκπρόσωπός της, στην απάντηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτείνει στο Κοινοβούλιο να αποφασίσει σχετικά με ψήφισμα που να καλεί τη Ρουμανία να λάβει τα απαραίτητα βήματα για να λάβει υπόψη τις, ε, τις ε, διατάξεις ε, της τις διατάξεις για την προστασία του παιδιού. Εγώ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρώ ότι αυτό είναι απαράδεκτη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι θέμα το οποίο θα παρακολουθήσω στενά και θα ρωτήσω στα ε, ανώτερα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν κάτι τέτοιο είναι ε, παραδεκτό. Αυτά είχα να πω. Κλείνοντας, παρακαλώ να κλείσετε την, ε, την αναφορά αυτή, διότι δεν υπάρχει καμία νομική βάση για την συζήτηση αυτή. Και δεν μπορεί εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθεί να μα επηρεάσει σχετικά με το ότι θα βάλουμε στη μέση διάταξη τη ε, της Επιτροπή μα. Ότι ήμουν στη θέση του νομοθέτη το 2001, αντιμέτωπη με αυτή την τραυματική εμπειρία στη Ρουμανία, ίσως ε, έκανα ακόμη και σκληρούς νόμους σε ό,τι αφορά την προσπάθεια να ανατρέψω το τράφικινγκ των παιδιών σε όλη αυτή τη διάρκεια. Επομένως θεωρώ ότι ήδη η Ρουμανία από το 2004 κάνει προσπάθεια να αναθεωρήσει από μόνη της τον, ε, του, τους όρους με βάση τους οποίους θα προχωρήσει σε μια διεύρυνση των όρων για, για την, ε, των, ε, των κριτηρίων για, τις, για την υιοθεσία. Εκτιμώ ωστόσο ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορέσει να συμβιβαστεί με μια νέα εικόνα και είναι υποχρεωμένη νομίζω η κυβέρνηση να προστατέψει τα παιδιά της. Θα έλεγα ότι η Ευρώπη έχει την υποχρέωση να καλύψει ένα κενό που αφορά στην υιοθεσία στην Ευρώπη και βεβαίως και ένα άλλο ακόμη πιο σημαντικό κενό να βρει τρόπους να ελέγξει τα αποτελέσματα αυτών των υιοθεσιών να παρακολουθεί δηλαδή τα παιδιά που κάποια στιγμή υιοθετήθηκαν και δεν ξέρουμε ή ξέρουμε πού βρίσκονται. Μέχρι ότου λοιπόν βρει ένα δίκαιο που δεν θα είναι απλώς διακρατικές συμφωνίες αλλά θα είναι ευρωπαϊκό δίκαιο για την υιοθεσία και θεωρώ τεράστιο κενό ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο, ένα. Και μέχρι ότου βρει τρόπους να κάνει follow-up σε αυτές τις υιοθεσίε, η Ρουμανία μπορεί να κάνει αυτό που εκτιμά και αυτό που όλοι μα θεωρούμε ότι κάνει σωστά. Να προστατέψει τα παιδιά της μέχρι ότου διασφαλίσει απολύτως το μέλλον τους. Ε, Ο κύριος Κάσμαν, αλλά πριν του δώσω το λόγο, να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε ελάχιστα λεφτά μόνο στη διάθεσή μας, γιατί σε λίγο, στις 6.30 δηλαδή, θα σταματήσει η διερμηνία. Άλλωστε έχουμε και αύριο, και αύριο μέρα είναι. Κύριε Κάσμαν, παρακαλώ χρόνου φίδου. Θα είναι η τελευταία παρέμβαση τη ημέρα, γιατί περιμένουμε και την απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Κάσμα. Uh, Κυρία Πρόεδρε, όσο λιγότερο συζητάμε την ε, πίεση του χρόνου, τόσο περισσότερο χρόνο έχουμε να μιλήσουμε. περιπτώσει, εγώ είμαι υπεύθυνο για το μορατόριο. Εγώ ήμουν εισηγητή για τη Ρουμανία των, ε, των Σοσιαλιστών. Ε, συνεργάστηκα στενά με την Βαρόνι Νίκολσον και εμεί και οι, κυρί, οι κύριε πολιτικέ ομάδε του Κοινοβουλίου ζήτησαν να δοθεί τέλος ε, στο, στο καθεστώς διεθνών υιοθεσιών. Εμείς ζητήσαμε το μορατόριο. Δεν συμφωνώ ότι υπάρχει βάση να προχωρήσουμε. Σίγουρα δεν υπάρχει νομική βάση και σίγουρα δεν υπάρχει λόγος ε, να επικαλεστούμε το άρθρο 7. Επιτρέψτε μόνο να πω, ήταν έντονη η συζήτηση. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει ε, παραβίαση των συνθήκων. Θα έπρεπε εδώ να συζητάμε τα ε, δικαιώματα των παιδιών και την ευθύνη απέναντι στο παιδί. Εάν υπάρχουν προβλήματα για τα παιδιά στη Ρουμανία, δεν μπορούμε να εξάγουμε το πρόβλημα. Θα πρέπει να ζητήσουμε από κάθε χώρα να τηρήσει τι υποχρεώσει τη προ του ε, πολίτε τη συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Ξαφνικά, το να στέλνει κανεί για υιοθεσία ένα παιδί σε άλλη χώρα δεν πετυχαίνει τίποτα Ίσως μόνο για ένα παιδί, εντάξει, όσο καλό κι αν είναι αυτό. Αλλά εφόσον παρακολουθούνται τα παιδιά ε, μετά, δεν μπορούν όλα τα παιδιά να δοθούν ε, προς ε, διεθνή υιοθεσία και το μόνο πράγμα που ε, μας ενδιαφέρει εδώ είναι το δικαίωμα του παιδιού να έχει τους καλύτερους ε, θετούς γονείς. Κανένας Κανένα δεν έχει δικαίωμα να υιοθετήσει, αλλά έχει δικαίωμα να εξεταστεί. Ε, και η Ρουμανία μπορεί να λέει ότι εντάξει, ε, δεν πληρείται όμως τα, ε, προσόντα για, να γίνεται θετός γονιός. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σύστημα φροντίδα των παιδιών που υιοθετούνται εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά θα υπάρξουν εξελίξει, αλλά μία μη κυβερνητική οργάνωση από την Ιταλία κατά των ε, ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων και των Υπουργείων ε, τη Ρουμανία, που πιστεύουν ότι γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση και που στο κάτω-κάτω τη γραφή έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη του παιδιού. Θα πρέπει να σεβαστούμε λοιπόν τους ε, Ρουμάνους. Δεν έχει γίνει κανένα λάθος. Ε, ε, καλές προθέσεις υπήρχαν για να προστατευτούν τα δικαιώματα των παιδιών. Γι' αυτό καταλήγω στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να κλείσουμε την αναφορά αυτή. Ευχαριστώ. Grazie δεν ε, ζητάει κανένα άλλο συνάδελφο το λόγο. Κοιτάξτε, είμαστε στο όριο του χρόνου. Αν θέλουμε μπορούμε να συζητήσουμε τη συζήτηση αύριο, γιατί έχουμε φτάσει στις ή 6.30. Εκτό αν θέλουμε να συνεχίσουμε χωρί διερμηνεί, στα αγγλικά. Μπασινάρο. Κύριε Πρόεδρε. Εγώ είπα, αφού συζητήσουμε την αναφορά αυτή, να αποφασίσουμε, να ψηφίσουμε. Ή θα κλείσει η αναφορά ή θα παραμείνει ανοιχτή. Καλό να ψηφίσουμε να κλείσει η αναφορά αυτή. Πρόεδρος, συμφωνώ. Αυτό ακριβώ θα πρότεινα. Την πρότασή σας θα υπέβαλα. Αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε αύριο το πρωί αν θέλετε. Γιατί σήμερα δεν έχουμε χρόνο. Σίγουρα θα πάρω μια απόφαση. Αύριο το πρωί τρει συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Θα μιλήσουν. Θα μιλήσει και η τη Κομισιόν. Εσείς συνάδελφοι μπορείτε να ζητήσετε να ξαναμιλήσετε σε τέταρτο στη λίστα. Δεν έχουμε χρόνο. ένα μισή λεπτό μας μένει. Αύριο το πρωί. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Εκτός αν θέλετε να συνεχίσουμε σήμερα στα αγγλικά. Νομίζω σκοπιμότερο είναι να διακόψουμε για σήμερα και να συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 10 μετά τη συνάντηση των συντονιστών. Ci aggiorniamo allora domani mattina, grazie. Avrei το πρωί. Possinaro. Ok, Perché sono le 18.30. E Κοιτάξτε, είναι 6.30. Συνάδελφε, μιλήσαμε πρώτα, κάναμε τις αναφορές με τους αναφέροντες παρόντες. Το πρώτο, το ισπανικό, μας πήρε πάρα πολύ χρόνο.